I'm sorry, we have to start because we have... Να ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Τεσσερσήμιση, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε την συνεδρίαση αυτή. Θα ασχοληθούμε με το σημείο 11 τώρα, την εφαρμογή της οδηγίας 2008 κάθετο 48 για την καταναλωτική πίστη. Η ΕΚΟΝ θα γνωμοδοτήσει στην ΙΜΚΟ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ο Θείοντορ Στόλο Γιάννη είναι ο εισηγητής. Θέλω να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για σας για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταρχάς, ο εισηγητής είναι ο κύριος Λέχνερ, που υποτίθεται ότι θα φύγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε νέο εισηγητή και δεν έχουμε σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ετοίμασα την, το σχέδιο γνωμοδότησης χωρίς να έχω το σχέδιο έκθεσης. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες ε, δύο εργασίες ε, εν εξελίξη για το ίδιο θέμα. Για το άρθρο 27 της Οδηγίας ε, για την Καταναλωτική Πίστη. Η Κομισιόν θα κάνει κάθε πέντε χρόνια και για πρώτη φορά στις 12 Μαΐου 2013 μία αναθεώρηση αυτής της οδηγίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν του χρόνου θα κάνει μια πρόταση για το πώς θα αλλάξει αυτή η οδηγία. Και η Κοινή Επιτροπή των, αρχών, των εποπτικών αρχών θα υιοθετήσουν μια ενδιάμεση στρατηγική και μία ανάλυση για την προστασία των καταναλωτών, ούτω ώστε να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ε, διατομεακές. Υποτίθεται ότι θα είναι έτοιμη το πρώτο εξάμεινο του 2013. Τώρα, το θέμα μας, η καταναλωτική πίστη. Διευκολύνει την πρόσβαση σε ε, υπηρεσίες ε, όπως μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, οπτικοακουστικά, διάφορες υπηρεσίες, φοιτητικά δάνεια, είναι προσωπικά δάνεια, ε, πιστοτικές κάρτες, ε, δάνεια. Μιλάμε για πίστη, για καταναλωτική πίστη, για διάφορα θέματα, για αυτοκίνητα, που είναι 12.400 ε, ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ για άλλα θέματα αλλάζουν τα ποσά. έχουμε έρθει σε επαφή με ενώσεις και το σύνολο του ποσού της αγοράς είναι 1-3 ευρώ. Το σύνολο της καταναλωτικής πίστης που δίδεται. Υπάρχει μια μελέτη για αυτή την οδηγία της καταναλωτικής πίστης που βασίστηκε σε έρευνες ε, που έγιναν σε 14 κράτη-μέλη, τον τρόπο λέει, που εφάρμοσαν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η μεταφορά της οδηγίας είναι ικανοποιητική, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Καταρχάς, ίσως και πιο σημαντικό για μας, είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονταν, δεν ήταν η πρόθεση της οδηγίας να τα καλύψει, αλλά τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να τα καλύψουν με την εφαρμογή της οδηγίας. Ε, πιστοτικές συμφωνίες ε, για τα ε, ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ενυπόθηκα δάνεια, α, κινητή περιουσία κτλ. Επίσης, σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει κατόφλι ούτε ανώτατο όριο. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο 200 ευρώ και ένα μέγιστο όριο 75.000 ευρώ. Υπάρχει μόνο μία χώρα, η Αυστρία, όπου υπάρχει μία αναφορά για το, την κατανοητική πίστη σε ξένο συνάλλαγμα και στην πραγματικότητα πρόκειται για πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν στους καταναλωτές για τους κινδύνους ε, τέτοια πίστη σε ξένο συνάλλαγμα. Τι έχει εδώ πέρα το σχέδιο γνωμοδότησης. Λάβαμε υπόψη ότι η οδηγία για την καταναλωτική πίστη εκδόθηκε πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση. Η καταναλωτική πίστη ήταν λόγος που οδηγηθήκαμε στην κρίση. Και μάλιστα η κανονική πίστη σε ξένο συνάλλαγμα ήταν ένα κίνδυνο, μεγάλο σε Ουγγαρία, όπως η ε, Ουγγαρία, η Ρουμανία και άλλε χώρε που χρησιμοποίησαν πάρα πολύ αυτού του είδου την κανονική πίστη σε ξένο συνάλλαγμα. Υπάρχει και μία σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου τη 21 η Σεπτεμβρίου του 2011 για το δανεισμό σε ξένονομίσματα γενικά. Υπάρχει προτινόμενη σύσταση καταρχάς να δοθούν στους καταναλωτές παρκείς πληροφορίες για τους κινδύνους, για, σε αυτό τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα, σε όλες τις φάσεις, προσυμβατικά και στις ε, συμφωνίες τις πιστοτικές. Αυτή είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Το δεύτερο είναι δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα θα πρέπει να δίνονται μόνο σε καταναλωτέ που αποδεικνύουν την πιστοληπτική τους ικανότητα. Όπως είπα και πριν, υπάρχει μόνο μία χώρα που έβαλε στην εθνική της νομοθεσία πληροφο... κάποια υποχρέωση για πληροφορίες που να αφορούν τον κίνδυνο για τους καταναλωτές εφόσον δανείζονται σε ξενονόμισμα επίσης. Η τρίτη σύσταση αφορά τους όρους της καταναλωτικής πίστης. Και η προθεσμία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να δανειζόμαστε για πάνω από πέντε χρόνια. Γιατί Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα δάνεια αυτά τα κανονικά δίνονται για παραπάνω από 5 χρόνια, 7, 8 κτλ. Δεν μιλάμε τότε για κανονική πίστη αυτή καθεαυτή όταν ξεπερνάει την πενταετία. Η τέταρτη σύσταση είναι ότι δεν θα πρέπει η εγγύηση να είναι το σπίτι του καταναλωτή όταν έχουμε μόνο ένα μισθωτό στο νοικοκυριό. Βασικά. Και ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σύσταση. Γιατί στις πρώην ε, σοσιαλιστικές χώρες, όπου ο πληθυσμός δεν ήξερε πολλά από τη χρήση της πίστοσης των δανείων κτλ. Οι τράπεζες εγγυόνταν τα δάνεια που έδιναν στους καταναλωτές με ενυπόθηκα δάνεια, με το σπίτι τους. Και τώρα βλέπουμε καταναλωτές που κατέληξαν στο δρόμο, γιατί οι τράπεζες πουλάνε τα σπίτια τους, τα οποία έχουν κατασχέσει. Η τελευταία σύσταση είναι ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ ε, διαφόρων παρόχων και να αγοράσουν βοηθητικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη μια ασφάλεια. Συνήθως ε, συνδέονται αυτές, αυτή η καταναλωτική πίστη με ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Ε, τουλάχιστον αυτό ισχύει σε κάποιες χώρες. Σταματάω εδώ και θα ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Κυρία Σουίνμπεργκ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Χρειάστηκε να παρέμβετε καθοδόν, χωρίς να έχετε τη βασική έκθεση από τη Βασική Επιτροπή. Υποστηρίζω τις εκκλήσεις σας για θέματα που αφορούν το δανεισμό σε ξενονόμισμα και στη δική μου χώρα, ε, όπου θέματα της κανονικής πίστης ε, αφορά άτομα που έχουν και δεύτερα σπίτια. Παρ' όλα αυτά έχουμε εμπειρία ε, που ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους αυτού του δανεισμού. Ε, νομίζω ότι αυτό το θέμα δηλαδή αφορά πολλές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, καλό είναι που το θέτετε. Ένα-δύο σημεία είναι πολύ καλά και αφορούν πολλές χώρες. Ε, Επίση συμφωνώ ότι το νούμερο 5 ε, για την ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να διαιρούμε αυτές οι υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να συνδεθούν αυτές οι υπηρεσίες ε, με ασφαλιστικά προϊόντα. Θα πρέπει να συνδεθούν μάλλον συγγνώμη, με ασφαλιστικά προϊόντα. Όλα αυτά είναι καλά. Ε, χαίρομαι για τις εξηγήσεις που δώσατε για το νούμερο 3, γιατί δεν καταλάβαινα ακριβώς τον όριο αυτό που βάζατε τις πενταετίας. Δεν μπορούσα να φανταστώ προϊόντα πέραν της πενταετίας. Ε, μας εξηγήσατε ότι υπάρχουν προϊόντα σε άλλα κρατημέλη που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Μήπως θα μπορούσαμε να ορίσουμε, να τα δούμε αυτά τα προϊόντα και τι επίπτωση θα μπορούσε και να δούμε ε, τι θα σήμαινε αυτή η απαγόρευση του να ξεπεράσουμε την πενταετία. Τι εναλλακτικέ ε, υπάρχουν για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεπεράσουν την πενταετία. Επίσης, προσπαθώ να καταλάβω το νούμερο 4. Σε πολλές περιπτώσεις φαντάζομαι ότι οι οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν τέτοια πίστη μέσω διαφόρων συμβολέων και τα λοιπά, διαφόρων ρυθμίσεων. Ε, ξέρω ότι ας πούμε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην δική μου εκλογική περιφέρεια που έχουν ένα μισθό. Εάν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο, δεν θα αποκοπούν από την αγορά και δεν θα αναγκαστούν να πάνε σε τοκογλύφους, ε, σε παρόχους που δανείζουν με μεγάλο τόκο. Έχουμε πολλούς ε, οι οποίοι είναι πραγματικοί τοκογλύφοι και δίνουν τέτοια βραχυπρόθεσμα δάνεια στην Βρετανική αγορά. Ε, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υποθήκες ε, τα σπίτια τους, ε, μπορεί να αναγκαστούν να δανειστούν με τεράστια επιτόκια από παρόχους που δεν έχουν τόσο καλή θύμη, αν δεν τους εξασφαλίσετε και αυτή την εναλλακτική δυνατότητα. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και ίσως να δούμε πώς μπορούμε να το διατυπώσουμε, τόσο ώστε να μην εξαναγκάσουμε ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ε, πιο προβληματικές ε, πηγές για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Νομίζω ότι με το διάλογο μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια από τα θέματα και να καταλάβουμε ε, πώς λειτουργεί το πράγμα σε άλλες χώρες από τη δική μας. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε μπορώ να συμφωνήσω, μια και πρόκειται εδώ για τον τομέα όπου ζητείτε οι καταναλωτές για τους πιθανούς κινδύνους να μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα το τι θα συμβαίνει Υπάρχει το πρόβλημα των ταχαίων πιστώσεων στις αγορές και αυτό για πολλούς καταναλωτές στη χώρα μου είναι ένα μέσο το οποίο δεν κατανοούν και έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις για αυτούς. Δεν θα είχα τίποτα το αρνητικό να πω για το κείμενο κατά τα άλλα. Unfortunately, at least uh, I didn't get. Δεν είχα την διερμηνία των όσων είπατε και δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Θα το πω στα αγγλικά λοιπόν, ώστε να μην χρειάζεται να περιμένετε. Είναι θετικό λοιπόν θα έλεγα, ένα θετικό έγγραφο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και το υποστηρίζω απόλυτα. Ιδιαίτερα όπως για την, πρόταση, την πρώτη πρόταση ότι πρέπει να διευρυνθεί η γνώση των καταναλωτών για τους κινδύνους που συνεπάγονται τέτοια δάνεια πολλοί νέοι, ιδιαίτερα στην Φινλανδία, έχουν αρνητικά βιώματα, αρνητική πείρα όταν έχουμε τέτοιου είδους βραχυπρόθεσμα δάνεια και ε, όταν με αυτά τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ξεπερνούν τα, τους δικούς τους πόρους και δυνατότητες. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω, υποστηρίζω το έγγραφο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίγκολτ και μετά ο κύριος Σμιτ παρακαλώ. Κύριε Γκίγκολτ, έχετε τον λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μπορώ να λάβω τον λόγο και να πω τις απόψεις μου σε σχέση με τη, και το θέμα αυτό πριν από την Άλντε. Κάποια σύντομα σχόλια. Ευχαριστούμε για το σχέδιο το οποίο μας υποβάλατε. Και θα ήθελα και κάποιες τροπολογίες επιπρόσθετα θα καταθέσουμε. Ένα θέμα είναι, αυτή τη στιγμή διαβουλευόμαστε για μια ειδική ξεχωριστή οδηγία για τις στεγαστικές υποθήκες που στο τέλος τέλος δεν έχει και τόσο πολύ ε, νόημα να έχουμε δύο διαφορετικές οδηγίες για το ίδιο θέμα, μόνο πολλαπλασιάζει τις οδηγίες μια κοινή οδηγία για αυτά τα δύο θέματα θα ήταν σωστή, όπου θα εξετάζονται ξεχωριστά κάποια πράγματα εκεί όπου υπάρχουν διαφορές. Αυτό θα κάλυπτε τις ανάγκες σε σχέση με τις επικαλύψεις ούτως ή άλλως και γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό βάρος, την γραφειοκρατική επιβάρηση, απαλήφωνοντας το ένα, τη την άλλη οδηγία μακροπρόθεσμα. Ε, το θέμα τίθεται γιατί έχουμε δύο οδηγίες, παρότι πολλοί ορισμοί προσδιορισμοί είναι ταυτόσιμοι. Ερώτημα, γιατί έχουμε λοιπόν δύο ξεχωριστές οδηγίες. Δεύτερο, το δεύτερο αφορά το ότι βλέπουμε ένα πρόβλημα να υφίσταται με τον τρόπο με τον οποίο το ετήσιο ποσοστό τελών η επιβάρυνσης καθορίζεται στην οδηγία για τους καταναλωτές και τα δάνεια. Ιδιαίτερα όταν έχουμε ξένες δάνεια σε ένα συνάλλαγμα, μπορεί αυτό να είναι παραπλανητικό, διότι το APR υπολογίζεται μόνο στα πολύ πρόσφατα γεγονότα, ενώ μπορεί να υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στο μέλλον, οι διακυμάνσεις. Και αυτό ε, δίνει κίνητρα ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο στο οποίο όμως μπορεί να υπερχρεώνονται οι καταναλωτές. Γι' αυτό ακριβώς ε, σε σχέση με το πλαίσιο της οδηγίας θα υποστηρίζαμε να ληφθεί υπόψη η πρόταση ότι θα πρέπει να ενημερώνονται οι καταναλωτές δίνοντας τα απόλυτα μεγέθη και αριθμούς των μηνιαίων πληρωμών, μηνιαίων πληρωμών ή καταβολών που θα ήταν η συνέπεια συγκεκριμένων συμβάσεων. Διακόπτεται ο μιλητής χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση, δεν ακούστηκε. Περιμένω μέχρι να σταματήσει αυτή η φασαρία και ο θόρυβος. Παρακαλώ σταματήστε τις συνομιλίες εκεί. Προσέξτε, σταματήστε. Yeah, yeah, One after the other. Ναι, ο ένας μετά τον άλλο, το ένα μετά το άλλο. Εντάξει, λοιπόν, το πώς το APR υπολογίζεται θα μπορούσε να βελτιωθεί για τους καταναλωτές δίνοντας σε απόλυτα μεγέθη τις ε, μηνιαίες ε, πληρωμές ε, που πρέπει να γίνονται ας το πούμε έτσι μεταξύ του ελάχιστου και του, του μεγίστου ποσού που θα μπορούσε να συνεπάγεται μια συγκεκριμένη σύμβαση, ένα συμβόλαιο. Και θα πρέπει το μέγιστο να είναι το ανώτατο ανώφλιο, ώστε να είναι διαφανές για τον καταναλωτή ποια θα είναι η μέγιστη πληρωμή, η μέγιστη καταβολή μηνιαία και ποιες επιπτώσεις θα είχε αυτή η σύμβαση. Θα υπήρχε απόλυτη ελευθερία συμβατική ούτως ή άλλως, αλλά θα είχαμε απόλυτη διαφάνεια ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να το δουν αυτό. Ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες, επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης σύμβασης ενός συμβολέου και νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν μια σαφής βελτίωση αν μπορούσε να γίνει και θα καταθέσουμε αντίστοιχα τροπολογίες από πλευρά μας. Το πώς υπολογίζεται το APR πρέπει να αλλάξει και σε μηνιαίες καταβολές ή ε, πληρωμές θα πρέπει να ενημερώνονται τι θα πρέπει να πληρώνουν οι καταναλωτές έχοντας και το ανώτατο κατόφλιο ταυτόχρονα που θα γνωρίζουν ποιο θα είναι ώστε εκείνοι οι οποίοι θα προσφέρουν πιστώσεις και δάνεια να μπορούν να αποφασίζουν ποιο θα είναι το μέγιστο ποσό σύμφωνα με τις αλλαγές που μπορεί να επέρθουν λόγω των διακοιμάσεων των ισοτιμιών, των συναλλαγματικών ισοτιμιών κτλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψη του κυρίου Ντεμπάκερ όπως σας την παρουσιάζω. Θέλει να σας ευχαριστήσει για το σχέδιο που παρουσιάσατε σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Το μόνο έγγραφο το οποίο είναι διαθέσιμο είναι η μελέτη του Ιανουαρίου 2012 από την, ε, το τμήμα πολιτικής ε, είναι όμως ενδιαφέρον αυτό. Παρόλα αυτά δεν θα έπρεπε στην γνωμοδότηση να αναφέρουμε κάποια, ε, κάποιες από τις τράπεζες που καλυπτόντουσαν από αυτή τη μελέτη. Παρότι η μελέτη ήταν για την ΙΝΚΟ Πιστεύει ο κύριο Ντεμπάκερ ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιε πτυχέ αυτής της μελέτης στη γνωμοδότηση τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να υπάρξει περαιτέρω μελέτη για αυτέ τι ε, ε, εφαρμογέ και τι επιπτώσει του, Πρώτον, θα ήθελε να γνωρίζει ποιο είναι το κόστο του CCED στην εφαρμογή. Το κόστος αντανακλάται σε σχέση με το κόστος των, στους καταναλωτές. Δεύτερη ερώτηση η CCI, Standard European Credit Information Sheet, οδήγησε στο να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και γνώση από πλευράς των καταναλωτών για αυτά τα θέματα. Τρίτο ερώτημα. Υπάρχουν περισσότερα τέτοια δάνεια και πιστώσεις διασυνοριακά χάρη, χάρη σε αυτή την CCD. Έχει κάποιες ερωτήσεις λοιπόν ο κύριος Ντεμπάκερ προτείνει ο εισηγητής να μην υπάρχει μεγαλύτερο πλαίσιο από πέντε έτη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των καταναλωτών και των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Διαφορετικά θα έχουμε υψηλότερες πληρωμές και αυτό θα είναι διαθέσιμο μόνο για πλουσιότερους, ιδιαίτερα όσον αφορά το μέγιστο ποσό 75.000 ευρώ για ε, πιστοτική τέτοια ε, υπόθεση που είναι αδύνατο να αποσβεστεί, να ξεπληρωθεί σε πέντε χρόνια. Για τη δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο εδάφιο, θα πρέπει να γνωρίζουν πώς μελλοντικά θα διακυμένονται οι, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για να μπορέσουν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις. Αυτό είναι ανέφικτο. Αλλά και στην παράγραφο τέσσερα υπάρχουν προβλήματα. Πρώτα απ' όλα θα διασφαλίζεται το, η πίστοση ώστε να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών σε σχέση με τις, τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεύτερον, δεν είναι εύθετο να υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση για τις οικογένειες που έχουν μόνο έναν εργαζόμενο, έναν μισθωτό, ο οποίος συνεισφέρει ε, στα έξοδα του νοικοκυριού. Ο κύριος Ντεμπάκερ πιστεύει ότι πολλή δουλειά πρέπει να γίνει σε αυτό το σχέδιο και προσβλέπει να συνεργαστεί μαζί σας το επόμενο διάστημα τις επόμενες εβδομάδες. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσουμε εδώ πέρα τη συζήτηση. Προθεσμία για τροπολογίες. Δεν ναι, θα κάνω κάποια σχόλια, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω τα διαδικαστικά. 12 Απριλίου λοιπόν για τις τροπολογίες, η εξέτασή τους 7 Μαΐου. 12 Απριλίου λοιπόν για την κατάθεση των τροπολογιών. Να σας πω κάποια πράγματα τώρα. Κύριε Κέι, συμφωνώ μαζί σας για τους κινδύνους της ε, σύστασης υπαριθμών 4 για τον ένα μισθό, τα νοικοκυριά με ένα μισθό και το τι θα γίνει. Μάλιστα με εντυπωσίασαν οι περιπτώσεις που είδα ε, οικογένειες που έμειναν στο δρόμο γιατί οι τράπεζες ε, τους κατέσχεσαν τα σπίτια. Αυτό μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το σταματήσω, αλλά βεβαίως ε, να συζητήσω μαζί σας πώς θα βρούμε μια λύση. Όσον αφορά κύριε Σμιτ τον όρο Μπορούμε να το συζητήσουμε και συμφωνώ μαζί σας πως ε, κάποιες συστάσεις από τη μελέτη μπορούν να μπουν στη γνωμοδότηση, αλλά κατά κάποιον τρόπο περίμενα ο εισηγητής ε, να λάβει υπόψη του αυτές τις ε, συστάσεις, αλλά μπορεί να γίνει, καθώς δεν έχουμε μέχρι τώρα σχέδιο έκθεσης και συμφωνώ και με τον κύριο Γκίγκολτ πως ο υπολογισμός του, της αλλαγής του επιτοκίου είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να φέρει μια μελέτη. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει αυτή τη μελέτη του χρόνου. Επόμενη συνεδρίαση 5η 12 Απριλίου 2012, 9 με 12.30. Κυρία Κέι, παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Ε, εμείς ως ε, μικρή ομάδα έχουμε πάρα πολλή δουλειά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες και αναρωτιέμαι, υπάρχει λόγος που βιαζόμαστε τόσο πολύ, μήπως να επεκτείνουμε λίγο την προθεσμία για τροπολογίες, μιας που δεν έχουμε και την ε, έκθεση, ούτως ή άλλως από την ε, κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή. Okay. Now it's a break. Μάλιστα, διακόπτουμε λέει ο πρόεδρος μέχρι τις 5.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 So, Ησυχία παρακαλώ. Είμαι σίγουρη πως έχετε πολλές ερωτήσεις, οπότε όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο το καλύτερο. Καλώς ήρθατε. αυτά βεβαίως τα διαδικαστικά. Έγκριση ημερήσια διάταξης δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσει ούτε ανακοινώσει τη Προέδρου υπάρχουν, οπότε περνάμε κατευθείαν στην ανταλλαγή απόψεων ε, τη ε, Τρόικας ε, με τις Επιτροπές Οικονομικής και Νομισματική Πολιτικής και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Βλέπετε πώς προεδρεύω εγώ και υπερβάμεις από την κάθε επιτροπή. Αντιστοίχω, ορίζω τον Όλη Ρεν, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και Αρμόδια για το ευρώ, τον Γιώργ Γκράσμουσεν μέλο του ΔΣ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Πολ Τόμσεν, αναπληρωτή διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επικεφαλής αποστολής για την Ελλάδα και βεβαίως τους βουλευτές. Το έργο της Τρόικας μία και εμένα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Βεβαίως αυτό δεν ήταν στόχος της Τρόικας, αλλά ήταν κάτι το οποίο παρατηρήσαν πως συμβαίνει με τόση κάλυψη από τα μέσα. Οπότε Καταληφθήκαμε την ευκαιρία να προσκαλέσουμε την ε, Τρόικα σε μια δημόσια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη των Επιτροπών που θα συντελέσει στην ενημέρωση του κοινού και στην αντίληψη των ε, στόχων του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας και των πιθανών συνεπειών. Έτσι αυξάνουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ε, Τρόικας. Ο χρόνος πιέζει θα ζητήσω λοιπόν από τους ομιλητέ να τοποθετηθούν αρχικά για 10 λεπτά και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσει και απαντήσεις ε, όπου θα είμαι πολύ αυστηρή με τους βουλευτές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τον λόγο έχει ο κύριος Ολυρέν. Σε ευχαριστώ Σάρων, αγαπητοί Περβάνς, κυρίε και κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις για την Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω και για τις ερωτήσεις που είχατε υποβάλει εκ των προτέρων, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, στις οποίες στείλαμε γραπτές ε, απαντήσεις Αποκινούμε τον Γιώργο Άσμουσεν της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι θα είναι σύντομη η εισαγωγή μου. Η κρίση στην Ελλάδα είναι μια τεράστια πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η κληρονομιά ετών ε, ανεύθυνων πολιτικών και χάρη στην ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ε, αποφύγαμε τα χειρότερα, μια κοινωνική καταστροφή. Αλλά είναι σαφές πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη στην Ελλάδα, ειδικά για τις ε, πιο ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Το έργο της ε, Κομισιόν και τολμώ να πω ολόκληρης της ε, Τρόικα εστιάζεται στο να βοηθήσει την Ελλάδα να αναδιαρθρώσει και να εξισορροπήσει την οικονομία της αυξάνοντας τις μεσοπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης. Τονίζω αυτές τις λέξεις, απασχόλησης και ανάπτυξης, αυτή είναι η βασική στόχη του προγράμματος ε, οικονομικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας. Μετά από τις ε, τεράστιες ανισορροπίες, η απαραίτητη προσαρμογή θα χρειαστεί χρόνο. Όμως δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις για το ότι δεν θα υπάρξει ούτε ανάπτυξη ούτε νέες θέσεις εργασίας χωρίς διόρθωση των οικονομικών ανισορροπιών να υπενθυμίσουμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά και γιατί είμαστε εδώ. Δεν θα γινόταν σήμερα αυτή η ακρόαση αν οι πολιτικές διαδοχικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα δεν είχαν οδηγήσει σε μη βιώσιμες ε, ανισορροπίες ε, απώλειες ανταγωνιστικότητας και πάρα πολλά ελλείμματα. Να αναφέρω κάποια νούμερα. Το 2008 η Ελλάδα είχε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 18% του ΑΕΠ. Το 2009 ένα δημοσιονομικό έλλειμμα σχεδόν 16% του ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα αυτού η Ελλάδα και ίσως και η Ευρωζώνη στο σύνολό της ήταν στο χείλος της καταστροφής το γεγονός αυτό και η πιθανή άτακτη χρεοκοπία όθησε την Ελλάδα να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τους εταίρους της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Απρίλιο του 2010. Έκτοτε, μετά από το αίτημα της Ελλάδας, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δονοτού από κοινού ως Τρόικα βοήθησαν την Ελλάδα να φέρει την οικονομία της σε μια πορεία βιώσιμη μαζί με το ΔΝΤ τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν ε, δεσμεύσει χρηματοδότηση 260 δισεκατομμυρίων ευρώ, άλλα 100 δισεκατομμύρια από πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, μέσω της ανταλλαγής που μειώνει την ονομαστική αξία των ομολόγων τους κατά 53,5%. Ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος και της χρηματοδότησης η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μειώσει το χρέος της από 160% σε 116% του ΑΕΠ το 2020, μια ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί. Η άνευ προηγουμένου οικονομική αλληλεγγύη που δόθηκε στην Ελλάδα αποδεικνύει πως υπάρχει μια ισχυρή πολιτική δέσμευση από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της ε, Ευρωζώνης για να δοθεί στην Ελλάδα ο χρόνος και τα μέσα να επανορθώσει τη ζημιά και να θεραπεύσει τα οικονομικά της προβλήματα. Και δεν είναι σωστό ούτε δίκαιο να κατηγορούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτούς που ήρθαν να βοηθήσουν αφού είχε γίνει ζημιά. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα. Η Κομισιόν αναγνώρισε δημοσίω πω η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλε δημοσιονομικέ προσαρμογέ υπό εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε. Αναγνωρίζοντας αυτές τις ε, προσπάθειες, ε, η Τρόικα συνέχισε να στηρίζει την Ελλάδα παρά το ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2010 και 2011 δεν είχαν επιτευχθεί πλήρως. Επίσης, αναγνωρίζοντας αυτές τις προσπάθειες, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν να αυξήσουν και να επεκτείνουν χρονικά την οικονομική στήριξη της Ελλάδας. Προκλήσεις παραμένουν. Ο ρυθμός προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων δεν είναι επαρκής για να καταστούν τα δημοσιοοικονομικά της Ελλάδας βιώσιμα ή για να κλείσει το κενό της ανταγωνιστικότητας άρα απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Η ομάδα η αρμόδια για την Ελλάδα είναι μια βοήθεια την οποία παρέχει η Κομισιόν στις αρχές Ελλάδας καθώς θέλουν να οικοδομήσουν μια σύγχρονη Ελλάδα με ευημερία. Πρόκειται για τεχνική αρρωγή η ομάδα αυτή δράσης των διοικήσεων των κρατών μελών προς την Ελλάδα για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που χρειάζονται για μια υγιή και στιβαρή ανάκαμψη. Ως αποτέλεσμα στοχεύουμε οι Έλληνες πολίτες να έχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίε, ένα αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα και ένα καλύτερο περιβάλλον για το επιχειρήν και τις επενδύσεις το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα έχει στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη, παραδείγματο χάρη οι περικοπές στις συντάξεις στόχευσαν τις υψηλότερες ε, συντάξεις και προστάτευσαν τις χαμηλότερες. Οι μειώσεις στο σύστημα υγείας είχαν στόχο να βελτιώσουν τις παροχές για τον απλό πολίτη και σημαντικότερο η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής παίζει κρίσιμο ρόλο για το πρόγραμμα όχι μόνο λόγω των εσόδων αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και αποδοχής του προγράμματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και πρέπει να της δώσουμε την ευκαιρία να το εφαρμόσει. Το πρώτο πρόγραμμα για την Ελλάδα μας διδάσκει ένα σημαντικό μάθημα. Είχε δύο αχίλιες φτέρνες. Η πρώτη ήταν η χαμηλή διοικητική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης η οποία δεν επέτρεψε να γίνουν όπως έπρεπε οι μεταρρυθμίσεις. Η άλλη ήταν η έλλειψη της απαραίτητης πολιτικής ενότητας που απαιτείται για να κινητοποιηθεί επαρκής στήριξη για απαιτητικές μεταρρυθμίσεις. Για το δεύτερο πρόγραμμα κινητοποιούμε όλη την βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στην ελληνική διοίκηση για να ενισχυθεί η ικανότητά της. Αλλά η άλλη αχίλιος τέρνα, η έλλειψη πολιτικής ενότητας, παρά το ότι βελτιώθηκε πρόσφατα, μπορεί να θεραπευτεί μόνο από τους Έλληνες πολίτες την ελληνική κοινωνία την ίδια. Οπότε, κυρίες και κύριοι, Λίγα λόγια για το πρόγραμμα και το πώς το αισθάνονται οι Έλληνες. Είναι ένα πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας και ανήκει στην Ελλάδα. Η Τρόικα βοήθησε στον σχεδιασμό του και ε, επιφορτίστηκε από τους πίστοτες, δηλαδή η Ευρωζώνη και το δόνο του και τους ε, φορολογόμενούς τους εμέσως να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος για λογαριασμό όσων χρηματοδοτούν το ελληνικό κράτος με ποσά τεράστια. Με άλλα λόγια, η Τρόικα μπορεί να διευκολύνει, να στηρίξει, αλλά σε τελική ανάλυση οι ίδιοι Έλληνες θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να μεταρρυθμίσουν τη χώρα τους και να έχουν την ευθύνη για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρονικό όριο. Ο Γιώργ Άσμουσεν έχει το λόγο τώρα. Θα ήθελα σας παρακαλώ η φωτογράφη να μην στέκεστε μπροστά στο Προεδρείο. Ε, υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θέλουν να δουν τους ομιλητές. Ε, παρακαλώ να είσαστε στους διαδρόμους ε, γιατί αλλιώς θα αναγκαστώ να σας ε, στείλω έξω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, με μεγάλη χαρά. Είμαι εδώ ενώπιόν σας μαζί με τους συναδέλφους και φίλους, με τον Πολ, με τον Όλη. Νομίζω η προσπάθεια οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας ε, είναι επώδυνη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι πώς η Ελλάδα έφτασε σε αυτήν την κατάσταση. Και ποια είναι η εναλλακτική λύση τώρα. Η βασική επίπτωση της ε, προσαρμογής ε, αντικανοτοπτρίζει τη σοβαρότητα των μακροοικονομικών ανισορροπιών που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών στην Ελλάδα. Οι δημοσιονομικές πολιτικές που ήταν λαθασμένες, η έλλειψη των διαφορετικών ε, μεταρρυθμίσεων, οι πολιτικές αυτές υπέσκαψαν την βιωσιμότητα του κρατικού χρέους και δημιούργησαν ένα τεράστιο χάσμα ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραμμα προσαρμογής δεν είναι αυτό που προκαλεί την ε, συρρήκνωση, την πρόσφατη συρρήκνωση του ΑΕΠ. Η σημερινή οικονομική κατάσταση είναι μια αναπόφευκτη διόρθωση του προβλήματος που έχει συσσωρευτεί και δημιουργηθεί μέχρι το 2009. Υπάρχει εναλλακτική στο τρέχον πρόγραμμα προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Νομίζουμε ότι δεν βοηθούμε την Ελλάδα, δημιουργούμε ψεύδεις προσδοκίες. Οι εκκλήσεις για να χαλαρώσουν τα, δημοσιονομικά πρότυπα είναι αυταπάτη. Ε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικά προβλήματα. Δεν έχει πρόσβαση στις αγορές και μόνο μπορεί να υποφεληθεί από την επίσημη οικονομική βοήθεια που τη δίνουμε. Υπάρχει μόνο ένα δρόμο προ τα εμπρό, να αποκατασταθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα και με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθει η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιμείνει η Ελλάδα για να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση και να εφαρμοστούν ε, συνολικές διορθωτικές μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπιστούν επίσης οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα της Ελλάδας. Οι προσπάθειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και οι θυσίες ε, του ελληνικού λαού μέχρι στιγμής ήταν ουσιαστικές. Αλλά όμως ε, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Δεν είναι μυστικό ότι το πρόγραμμα υπόκειται σε απίστευτους κινδύνους ε, εφαρμογής. Η διαδικασία PCI, ε, PSI ήταν ε, ικανοποιητική και έχει βελτιωθεί ε, η βιωσιμότητα του χρέους. Μπορεί έτσι να φτάσει στο 116,5% το 2020 το χρέος. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει 100% το πρόγραμμα η δυναμική του χρέους είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε προβλήματα και βιολιστήσεις της εφαρμογής. Η δημοσιονομική εξυγίανση, η διαδικασία ε, ιδιωτικοποίησεων, οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, ε, θα, αν δεν συνεχιστούν, ε, δεν θα ε, υπάρξει ούτε ανάπτυξη, ούτε βιωσιμότητα. Θα έρθω να σταθώ σε τρεις τομείς. Ε, δημοσιονομική προσαρμογή, ε, ανταγωνιστικότητα και δημοσιονομικά θέματα. Για τη δημοσιονομική προσαρμογή, οι ελληνικές αρχές και ο ελληνικός λαός αξίζουν την αναγνώριση για τις ε, σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε δημοσιονομικό επίπεδο που κάναν τα τελευταία δύο χρόνια. Παρά την ύφεση, το κρατικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 6,5% του ΑΕΠ από το 2009 μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι από το 16% έφτασε σχεδόν στο 9%. Το μέγεθος ε, της ε, κυβέρνησης του δημόσιου τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το δυναμικό της Ελλάδας να εισπράξει. Επίσης, ε, η ποιότητα των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων δεν ήταν απόλυτα θετική. Ξεκίνησαν οι μεταρρυθμίσεις από τη μία, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο των μισθών του δημοσίου, ε, και το μη βιώσιμο επίπεδο των συντάξεων. Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις αυτές μέχρι στιγμής βασίστηκαν κυρίως σε αύξηση των φόρων ε, και σε γενικές μειώσεις των δαπανών. Κοιτώντας προς τα εμπρός, ε, η περαιτέρω πρόοδος σημαίνει εφαρμογή δύσκολων διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Το να κλείσει το χάσμα κατά 5,5% του ε, ελλείμματος ε, το 2013 και 2014. Αυτό θα είναι διαλήθος δηλαδή για την επιτυχία του προγράμματος. Χωρίς την θέληση της κυβέρνησης να σχεδιάσει και να εφαρμόσει αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις, τέτοιες μεγάλες προσαρμογές ε, δεν μπορούν να επιτευχθούν. Θα ζητήσω από την πολιτική τάξη της Ελλάδας να προχωρήσει παραβλέποντας τα συμφέροντα. Αλλιώς οι απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί αυτό το δημοσιονομικό χάσμα ε, δεν θα αποδώσουν. Ο Όλη μίλησε επίσης για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές προσαρμογές και το βάρος αυτών ε, κατανέμεται δίκαια. Ο βασικός τρόπος είναι μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Δυστυχώς μέχρι στιγμής η πρόοδος ήταν απογοητευτική σε πολλές περιπτώσεις οι πλούσιοι Έλληνες ε, συνεισφέρουν πολύ λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε στην προσπάθεια λόγω της φοροδιαφυγής. Η ενίσχυση της ε, διαχείρισης των, ε, του εισπρακτικού μηχανισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι μόνο χρειάζεται για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, αλλά θα βοηθήσουν για να γίνει αποδεκτό και κοινωνικά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, για την ανταγωνιστικότητα. Ε, υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα ήδη από το πρώτο πρόγραμμα, αλλά δεν ε, επετεύχθη αυτό που χρειάζεται. Ήδη η Ελλάδα ακόμα έχει ιστερεί ε, σε σχέση με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ε, μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει να κλείσει αυτό το χάσμα παραμένοντας η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά αυτό θα απαιτήσει πιο μεγάλη ε, εσωτερική υποτίμηση. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την δραματική αύξηση της ανεργίας. Θα πρέπει να μειωθούν οι ελάχιστοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα για μια στατηγική επιταχυμένης εσωτερικής υποτίμησης ε, εντός της Ευρωζώνης. Ίσως να μην είναι δημοφιλή αυτά τα μέτρα, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να τα αποφύγουμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τη βάση για ανανεωμένη ανταγωνιστικότητα και αύξηση της απασχόλησης. Δεν είναι ο μόνο τομέα όπου αποφασιστική δράση είναι απαραίτητη. Οι μεταρρυθμίσει τη αγορά-εργασία πρέπει να συμπληρωθούν από μια απελευθέρωση προϊόντων και υπηρεσιών, παραδείγματο χάρη τα κλειστά επαγγέλματα θα πρέπει να ανοίξουν. Η πολιτική βούληση είναι βασικό στοιχείο για να ε, ξεπεράσουμε τις ε, αντιδράσεις που υπάρχουν από διάφορα συμφέροντα. Επίσης, ε, τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση. Η Ελλάδα χρειάζεται κατεπηγόντως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραπεζικού τομέα. Ως συνέπεια του PSI, περισσότερες τράπεζες δεν έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση. Το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι τράπεζες οι οποίες είναι βιώσιμες και τις εκτιμάει έτσι η Τράπεζα της Ελλάδο θα ανακεφαλαιοποιηθούν. Ε, και όσες δεν μπορούν να αντλήσουν πόρους από την αγορά ε, θα αντλήσουν πόρους από αλλού. Οι τράπεζε που δεν είναι βιώσιμε θα πρέπει να εξηγιανθούν, θα πρέπει να κλείσουν. Τα 25 δις ευρώ ε, που δόθηκαν με την πρώτη εκταμείευση θα χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη ε, έγχυση ε, ρευστού στις ελληνικές τράπεζες. Το συνολικό ποσό για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι 50 δις ευρώ. Και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, δίδοντας ένα μήνυμα ελπίδας. Ναι, το φάρμακο είναι πάρα πολύ πικρό, αλλά ο ασθενής μπορεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του εάν ακολουθεί τη συνταγή του γιατρού. Κοιτώντας τις επιτυχείς παρελθούσες εμπειρίες δημοσιονομικής προσαρμογής και προσαρμογή τη ανταγωνιστικότητα και ανάκτηση ανταγωνιστικότητα σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, ε, μα δείχνει ότι δεν είναι χαμένη η μάχη. Αλλά η προπόθεση είναι μια ε, ισχυρή πολιτική βούληση ο ελληνικός λαός δεν μεταρρυθμίζει την οικονομία του και το κράτος του για να ικανοποιήσει την Τρόικα, για να ευχαριστήσει την α ή χώρα της Ευρωζώνης. Περνάει από αυτή τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων για το δικό του το καλό. Και επομένως, η ισχυρή πολιτική βούληση ε, πρέπει να είναι αναμενόμενη και είναι κλειδί στην επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχετε τον λόγο εσείς κύριε Πορτόμψαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, ομιλήσω για τον ρόλο της Τρόικας στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σύντομο σχόλιο για το πρώτο πρόγραμμα. Ενώ σε κάποιους τομείς δεν είχαμε τα ε, ευταία αποτελέσματα, τώρα υπάρχει μία τάση εντός και εκτός Ελλάδας να αγνοούμε το ότι έκανε μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα με αυτό το πρόγραμμα. Κυρίως η Ελλάδα έκανε πολλά για να αποκαταστήσει τον έλεγχο των δημοσιονομικών της. Η μείωση όσον αφορά το χρέος από το 15,5% στα 9,5% του ΑΕΠ ως ποσοστό είναι εντυπωσιακό γεγονός. Λίγες χώρες κατάφεραν τέτοια πράγματα σε δύο χρόνια και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα αντίξων ανέμων και σημαντική συρρήκνωση της οικονομίας ταυτόχρονα. Και αυτή η προσαρμογή βασιζόταν σε πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία αναπόφευκτα απαιτούσαν σημαντικές θυσίε από τους Έλληνες πολίτες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αποκαθιστώντας αυτό, το ότι έκανε πολλά η Ελλάδα, έχει ακόμα πολύ δρόμο να καλύψει, αλλά πέτυχε πολλά η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πρώτου προγράμματος και την εφαρμογή του. Στρέφομαι λοιπόν σε αυτό το νέο πρόγραμμα τώρα και Διαφωνώ με όλους εκείνους που λένε το νέο πρόγραμμα είναι μόνο θέματα δημοσιονομικής αυστηρότητας. Επικεντρώνεται έντονα στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Αλλά ξεκινήσω με τα δημοσιονομικά. Από το 10% ε, περίπου ε, που έχουμε του ΑΕΠ βρίσκεται η Ελλάδα σε μια δύσκολη κατάσταση. Καμιά χώρα δεν θα μπορούσε να έχει μια αηφόρο ανάπτυξη με τέτοιου είδους ε, ποσοστό. Και γι' αυτό η μείωση των δαπανών θα πρέπει να παραμείνει ένας ε, κέριος στόχος των οικονομικών πολιτικών. Ωστόσο αυτό σίγουρα συμφωνούμε με εκείνους που λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν πλέον οι φόροι και η φορολογία ή να υπάρξουν 200 αυξήσεις των περικοπών όσον αφορά τις συντάξεις και τους μισθούς. Για να αναφέρω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σάσμουσεν, πρέπει να κάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικές η Ελλάδα. Για τα έσοδα αυτό σημαίνει κυρίως ότι η Ελλάδα πρέπει να σημειώσει πρόοδο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτή η διεργασία έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία του προγράμματος προσαρμογής. Είναι το κλειδί για την κοινωνική αποδοχή από τους πολίτες μακροπρόθεσμα αυτού του προγράμματος. Και πρέπει οι ευκατάστατοι να, να πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Αυτό είναι ένας τομέας όπου έχει απογοητεύσει μέχρι σήμερα και το ομολογούμε αυτό το πρόγραμμα και υπάρχει ένας κίνδυνος να αποτύχει το πρόγραμμα αν δεν βελτιώσουμε τις ε, επιδόσεις μας. Μπορώ να πάω τόσο μακριά και να πω ότι δεν μπορώ να δω πώς η Ελλάδα μπορεί να, δια... διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη στους πολίτες και να διασφαλίσει ταυτόχρονα την δημοσιονομική εξυγίαση χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής κυρίως. Όσον αφορά το θέμα των δαπανών, οι διαθωτικέ μεταρρυθμίσεις απαιτούν κυρίως ε, το να βελτιωθούν ε, οι κοινωνικές ε, μεταφορές του κονδυλίων. Να δει κανεί τώρα το τι συμβαίνει σε σχέση με το ε, χρέος, δύο τρίτα οφείλονταν στην αύξηση κοινωνικών τέτοιων μεταθέσεων μεταφορών και περίπου κατά το ίμιση των συνολικών δαπανών. Κατεπηγόντως πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί ώστε ότι οι κοινωνικές μεταφορές θα διοχετεύονται σε εκείνους που χρειάζονται άμεσα αυτή την υποστήριξη. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνει με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Άλλα πράγματα που πρέπει να τονιστούν όσον αφορά τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο νομικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, είναι η συρρήκνωση του κυβερνητικού, του ρόλου της κυβέρνησης και του δημοσίου. Υπερβολικά πολλοί απασχολούνται στο δημόσιο και πρέπει αυτό να συνεπάγεται την ρήξη με ταμπού όσον αφορά την ε, ε, διαδικασία αυτή. Διότι δεν είναι πλέον χρήσιμη όλη αυτή η δημόσια υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρχει αυτή η συνιστόσα. Κάποιες από τις άλλες μεταρρυθμίσεις που έχουν σπουδαιότητα για την μείωση αυτών των βαρών όσον αφορά τον τομέα της υγείας βρίσκονται, έχουν ήδη προχωρήσει. Άλλες βρίσκονται σε πρώιμη φάση. Για να απαντήσω ερωτήματα τα οποία διατυπώσατε, αυτό είναι ένας τομέας όπου πραγματικά δυσχερέστατες μεταρρυθμίσεις μας αναμένουν και θα πρέπει να αναμείνουμε σημαντική αντίσταση από δεδομένα συμφέροντα. Η επιτυχία δεν είναι διασφαλισμένη λοιπόν με κανένα τρόπο. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να δω δεδομένων των επιδόσεων της Ελλάδας για τα δημοσιονομικά και τον αγώνα που έχει δώσει το πώς μπορούμε να δούμε αυτές τις επιδόσεις και να συμπεράνει κανείς ότι δεν έχουν το σθένος οι κυβερνητικές αρχές να πετύχουν και δεν έχουν τη βούληση να το κάνουν. Λοιπόν, τώρα αστραφώ στο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης. Τι κάνει το πρόγραμμα για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Και εδώ σε σχέση με την ύφεση κατά τη διάρκεια του 2011 δεν είχαμε τους ευταίους στόχους, δεν υλοποιήθηκαν. Κυρίως επειδή δεν φτάσαμε στην κριτική μάζα μεταρρυθμίσεων, διαθωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να αλλάξει η πορεία των, της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Εδώ υπάρχουν ελλείψεις και εδώ έχουμε την κυριότερη πρόκληση που αναμένει την κυβέρνηση σε σχέση με το νέο πρόγραμμα, να αναζωογονηθούν αυτές οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει ανάπτυξη διατυπώθηκε ένα ερώτημα. Αν ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων μπορεί να επιταχύνει και να αυξήσει αυτή την πορεία. Αυτό πρέπει να ε, διασφαλιστεί Ωστόσο, δεν είναι μόνο από πλευράς κυβέρνησης που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να βοηθήσει η κυβέρνηση αυξάνοντας τις επενδύσεις, τις υποδομές και τα δίκτυα. Όμως δεν υπάρχουν κονδύλια για να γίνει αυτό, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει το κεφάλαιο για να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Γι' αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον ιδιωτικό τομέα ο τομέα των επενδύσεων, οι επενδύσει ε, και στι ε, υποδομέ και στα δίκτυα. Υπήρξε και μια ερώτηση αν ε, ταμείο ιδιωτικοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των, δημοσίων, των επενδύσεων. βρίσκουμε στο πρόγραμμα φιλόδοξους στόχους για την ιδιωτικοποίηση αν αυτά τα χρήματα προσδιοριστούν για άλλη χρήση θα ανοίξει μεγάλο κενό όσον αφορά ε, τη χρηματοδότηση από πλευράς του προγράμματος. Και μια και έχουμε πολύ φιλόδοξο πλαίσιο εδώ, δεν υπάρχουν ελπίδες να είμαστε πιο επιτυχείς αν αλλάξουμε αυτό το πρόγραμμα. Τι κάνει λοιπόν το πρόγραμμα για να δώσει προώθηση στις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης έχουμε εδώ ένα χάσμα 15% και για να ανακάμψει η ανάπτυξη πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Και όπως είπε ο κύριος Άσμουσεν, μια και η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωζώνης, μόνο η εσωτερική υποτίμηση μπορεί να βοηθήσει να τα καταφέρουμε. Η κύρια επικέντρωση των μεταρρυθμίσεων πρόσφατα ήταν στην αγορά εργασία για να διευκολυνθεί η πραγματική ευθυγράμμιση των μισθών με την παραγωγικότητα. Νομίζουμε αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα για να διασφαλίσουμε μια έγκαιρη αντίδραση και ανταπόκριση, ώστε να μπορέσει σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο να υπάρξει αντιστάθμιση μέσω της ε, ε, διεύρυνσης των εξαγωγών που θα σημειωθεί. Όμως ε, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της αγοράς εργασίας δεν επαρκούν. Και εδώ συμφωνώ σίγουρα με εκείνους που λένε ότι θα αποτύχει το πρόγραμμα αν ο κύριος διάβλος ε, για την προσαρμογή θα είναι η συρρήκνωση του ΑΕΠ και η συρρήκνωση των μισθών αποκλειστικά. Δηλαδή αν η προσαρμογή επιτευχθεί κάνοντας την Ελλάδα 200 Θα πρέπει η Ελλάδα να γίνει πιο παραγωγική με διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν το σημαντικό δυναμικό για την αύξηση παραγωγικότητας από πλευρά της Ελλάδας ώστε να υπάρξει τόνωση της ελληνικής οικονομίας και το πρόγραμμα εμπεριέχει πολλά μέσα για να επιτευχθεί αυτό. Ένα από αυτά είναι να διασφαλίσουμε την απελευθέρωση της αγοράς ε, υπηρεσιών και προϊόντων. Αυτό θα διασφαλίζει ότι η μείωση μισθών θα αντανακλάται με χαμηλότερες, σε χαμηλότερες τιμές και αυτό θα διασφαλίσει μια έγκαιρη ενωρίς ε, ανάκαμψη ε, που θα σημειωθεί. Μέτρα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ε, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το πρόγραμμα έχει πάρα πολλά τέτοια μέτρα είναι πλήρες τέτοιων μέτρων για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να αποκατασταθεί η ανάπτυξη ενώ οι αρχές ε, έχουν δεσμευτεί να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις σε, όλες αυτές τις, ε, σε όλους αυτούς τους τομείς, πολλοί άλλοι τομείς ε, πρέπει να μπορέσουν να ενταχθούν και να καλυφθούν. Και πάλι αυτός είναι ένας τομέας όπου θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση από συγκεκριμένα συμφέροντα, δομημένα συμφέροντα. Αυτό θα πρέπει να είναι η επικέντρωση της διαρκούς μεταρρύθμισης που θα πρέπει να συνεχιστεί και δεν υπάρχει κάποια πανάκια, δεν υπάρχει μια μαγική ράβδος με ένα, με ένα μόνο πρόγραμμα, με μία δράση για την αποκατάσταση της ανάπτυξης. Όλα αυτά τα μέτρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να δράσουν με μια συγκεκριμένη αλληλουχία. Σύντομα να σχολιάσω το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους, όπου βλέπουμε ότι μειώνεται ε, η ε, διάσταση αυτή, παρόλα αυτά θα είναι πάρα πολύ υψηλό το χρέος και μάλιστα μέχρι και την επόμενη δεκαετία. Υπάρχει πολύ στενό περιθώριο για ελιγμούς ε, και για πολύ μικρό περιθώριο για ε, θέματα ε, φορολογικής εξαίρεσης ή δημοσιονομικής παρέκκλησης. Γι' αυτό λέμε ότι το πρόγραμμα για την ανάλυση των, πτυχών αυτών δείχνει κάποιες, κάποια αρνητικά στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη η Ελλάδα και να εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμα για να είναι επιτυχής η διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε κι εσείς ε, το χρόνο που σας είχαμε δώσει. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της συνάντησής μας, ε, δηλαδή το τμήμα ερωτήσεων-απαντήσεων. Όπως είπε και η Sharon Bowles, πιεζόμαστε πολύ από το χρόνο. Θα ήθελα ο κάθε ένας να είναι αυτοπιθαρχημένος για να μην χρειαστεί εγώ να δράσω όπως ακριβώς η Τρόικα. Θα ξεκινήσουμε με τους πρώτους τέσσερις ομιλητές. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον Ζων Πολ Γκοζές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, επί δεκαετίες οι δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας ξεπέρασαν τα έσοδα από τη φορολογία, συσσωρεύθηκε το χρέος με δραματικό τρόπο, οι κυβερνήσεις δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το χρέος, οι κεφαλαίες έκλεισαν στην Ελλάδα και σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση που γνωρίζουμε. Περί, περί, περιτό είναι να σκιαγραφεί σε αυτόν τον πίνακα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να θέσω ε, μία ερώτηση στον κάθε ομιλητή. Στον κύριο ε, Άσμουσεν, ε, ο οποίος νομίζω βγήκε λίγο από την πεπατημένη τον ευχαριστώ για όσα είπε και δεδομένου της διατύπωσής του, της διαπίστωσής του, θέλω να μου πει πώς εκτιμά την ικανότητα της Ελλάδας, πολύ συγκεκριμένα, να μετασχηματιστεί ε, επαρκώς και εγκαίρως, ούτως ώστε να γίνει ανταγωνιστική, για να ξαναβρει την, την ανάπτυξη και να αποπληρώσει το χρέος. Εάν αποτύχει το πρόγραμμα, τι θα γίνει ή αν οι Έλληνες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν ε, εκλέξουν μια απαραίτητη δεν δώσουν ε, την απαραίτητη πλειοψηφία ε, σε πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν δεσμευτεί απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα. Έπειτα, η Τρόικα, κύριε Τόμσεν, έχει τα μέσα και την ικανότητα για να βοηθήσει την Ελλάδα στην προσπάθειά της. Και ποιο είναι το κυβερνητικό επίπεδο, ποιοι είναι οι συνομιλητές σας, ποιοι είναι οι ομόλογοι της Τρόικα ε, με τους οποίους πραγματικά συνομιλείτε. Κύριε Ρεν, επίσης, δεν συμφωνώ με την ανάλυση ότι η Ελλάδα έθεσε εν κινδύνο την Ευρωζώνη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα επεκταθώ. Γιατί οι υπηρεσίες σας ε, καταβάλουν τόση προσπάθεια για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την αποτυχία ε, Είχατε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ε, νομική προστασία των κρατών που βρίσκονται σε δυσκολία, ούτω ώστε σε δύο, τρία, τέσσερα χρονια να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα είμαστε σε θέση να δράσουμε εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων. Ε, δεν θέλουμε. Θέλουμε να επιτρέψουμε σε ένα κράτος που είναι σε δυσκολία να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Γι' αυτό θέλω να ε, μιλήσω. Η τρεις ε, ομιλητές εδώ της Τρόικα μου θυμίζουν το, το παράδειγμα με τους τρεις επιθήκους. Μην δεν ακούω, δεν μιλάω κτλ. Δεν ξέρω τίποτα. Μιλάτε για τη μείωση των μισθών, μιλάτε για τη μείωση των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών. Ε, δεν νομίζω ότι έχετε σκεφτεί τίποτα άλλο. Ε, στην, ε, ο πληθωρισμός ε, αντικαταστάθηκε από μαζική αύξηση των φόρων. Ε, μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, ε, συρρυκνώθηκε ε, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, εξαφανίστηκαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί πέντε χρόνια είναι σε ύφεση η Ελλάδα και, και λόγω της ύφεσης θα αυξηθεί με μηχανικό τρόπο το χρέος. Ο κύριος Άσμουσεν και ο κύριος Τόμσεν λένε ότι ίσως η Τρόικα έχει τελικά, μετά από ανάγνωση των, ε, των εκθέσεών της, ε, ίσως έχει αμφιβολήσει ότι είναι αποτελεσματική. Η ύφεση είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι είχαμε προβλέψει. Η εσωτερική υποτίμηση που χρειάζεται για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα ε, βραχυπρόθεσμα αρκεί. Επίσης, ε, η μείωση στο κόστος των μισθών ε, δεν νομίζω ότι θα είναι επιτυχής για να προωθήσει τους, ε, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Συμφωνείτε με αυτό? Αν θέλετε να αποκατασταθεί η δύναμη της χώρας, θα πρέπει να υπάρξει μια δημοσιονομική ε, εξυγίανση για την δημοσιονομική εξυγίαση ήταν πολύ στεναρή, αλλά ήταν πολύ αδύναμη στους άλλους τομείς, ε, στον κοινωνικό τομέα, ε, στο θέμα της ανάπτυξης. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση που έκανε ο Ζατ Κλοντ Γιούνκερ στο Eurogroup. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚΑ. Από την Επιτροπή Ομπλουά, ο Ζορς Πακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος της Κοινωνικής Επιτροπής Πολλά ακούσαμε για τα δημοσιονομικά. Ακούσαμε και πολλά για την εξοικονόμηση κονδυλίων. Δεν ακούσαμε όμως για την απασχόληση σε σχέση με το six-pack ήδη τα εξαπλά μέτρα είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Δεν είναι όμως η πλήρης απάντηση για τη σημερινή κατάσταση και επαναλαμβάνεται αυτή η επίκριση σχετικά αργά εφέτος υπήρξε αντίδραση και έγινε λόγος για ανάπτυξη και απασχόληση και αύξηση της απασχόλησης και με πολλές επιφυλάξεις και δισταγμούς και έτσι χάθηκε εμπιστοσύνη σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθήσατε να ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη των αγορών. Χάσατε όμως ε, την εμπιστοσύνη των λαών, των πολιτών και των νέων και έχουμε ποσοστό ανεργίας Κάποιοι κάνουν πραγματικά λόγο για μια χαμένη γενεά και αυτό είναι απαράδεκτο. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ αρνητική και το Ευρωκοινοβούλιο ήδη έγκαιρα, όπως προαναφέραμε, είπαμε ότι δεν επαρκεί η λιτότητα και η εξοικονομήση κονδυλίων και πρέπει νέα πράγματα να γίνουν, νέες αρμοδιότητες για τους νέους, μια ευκαιρία στους νέους που πρέπει να δοθεί. Προτάθηκε και η εγγύηση για τους νέους, όπου μετά από το αργότερο τέσσερις μήνες ένας νέος θα μπορεί να έχει μια πρόσθετη θέση κατάρτισης για να μπορέσει να απασχοληθεί. Τώρα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξέταση 8 χωρών χωρών και μεταξύ αυτών και την Ελλάδα και θα ήθελα να ρωτήσω Πώς έχει το πράγμα με την έκθεση τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς έχει η κατάσταση, ποια μέτρα μπορούν πρόθεσμα άμεσα να αναλυθούν, διότι πιέζει ο χρόνος. Τι γίνεται με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και με τις υποδομές, δηλαδή να υπάρξει ένα διπλό κέρδος, άμεσα όμως αν δράσουμε και δεύτερον μακροπρόθεσμα όσον αφορά χρηματοοικονομικά ε, οικονομικά προγράμματα και σχέδια, κυρίως όμως μέτρα για τους νέους, για τις, τους και την απασχόληση, διότι στην Ελλάδα ε, εγκαταλείπουν την Ελλάδα μεταναστεύουν οι νέοι Έλληνες και αυτό έχει πάρει δραματικές διαστάσεις. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή αυτής της τετράδας από την Επιτροπή Απασχόλησης από την Ομάδα Σοσιαλιστών, κυρία Σιλβάνα Ράπτη, δύο λεπτά. Σας καλωσορίζω στις ε, επιτροπές μας κύριοι και σας δείχνω αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα ευρώ. Έχει δύο όψεις όμως. Στη μία όψη είναι οι αριθμοί. Στην άλλη όψη είναι οι άνθρωποι. Στη μία όψη είναι η λιτότητα και οι περικοπές. Στην άλλη άποψη, στην άλλη επιφάνεια, είναι η απασχόληση. Βλέπουμε μέχρι τώρα να μιλάτε, να ενεργείτε, να προτείνετε λύσεις μόνον σε σχέση με τη λιτότητα και τις περικοπές. Δεν λαμβάνετε καθόλου υπόψη σας τους εργαζομένους. Χτες ο Υπουργός Εργασίας της Ελλάδας είπε ακόμη έναν αριθμό. 400.000 εργαζόμενοι δεν πληρώνονται διότι εργάζονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομική ασφυξία. Επίσης, χθες το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας έβγαλε την έκθεσή του για το πρώτο δίμηνο του 2012. Και ξέρετε τι διαπιστώνει. Διαπιστώνει ραγδαία επιδείνωση των όρων εργασίας. Διαπιστώνει ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έχουν μειωθεί κατά 20% διαπιστώνει ότι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και η εκπεριτροπής εργασίας έχουν διπλασιαστεί. Διαπιστώνει για μια ακόμη φορά ότι η ανεργία και ιδιαίτερη η ανεργία των νέων καλπάζει. Θα ήθελα να μου απαντήσετε ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να πάρετε ώστε να αναστείλετε αυτή την κατάσταση. Θέλω τέλος να ρωτήσω κάτι ακόμη. Μιλήσατε για ασθενή στον ασθενή, έρχεστε ως γιατρός και δίνετε ένα πακέτο λιτότητας. Όπως άλλοι δίνουν ένα πακέτο ασπιρίνης. Για κάθε νόσο. Δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι δίνετε το ίδιο πακέτο φαρμάκου, τη λιτότητα, και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και όλοι οι ασθενείς με το που αρχίζουν να παίρνουν τα χαπάκια της λιτότητας, αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Παρακαλώ θα ήθελα το σχολιασμό σας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στους τρεις καλεσμένους της ε, Τρόικα για τέσσερα λεφτά ο καθένας. Ο Επίτροπος, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Λιρέν, έχει το λόγο πρώτος. Let me thank you for very substantive debate and, uh, Ευχαριστώ για την ε, ουσιαστική συζήτηση και τις πολύ σκόπιμες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση που μου απευθύνθηκε από τον κύριο Γκοζές. που αφορά το κεφάλαιο 11. Ε, στα πλαίσια του 2 ΠΑΚ της χρεοκοπίας. Προφανώς συνδέεται με το θέμα της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα και πώς θα πρέπει να οργανωθεί σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του χρέους. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματά σας, τους λόγους, αντιρρήσεις σας. Θέλετε να προστατευτεί ο φορολογούμενος και να μειωθεί το άμεσο βάρος. Πρέπει να τονίσω όμως ένα τέτοιο θεσμοθεστημένο σύστημα εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα θα έχει αυτόματο χαρακτήρα ή μη αυτόματο χαρακτήρα μέσω της νομοθεσίας. Και αν ναι, θα είχαμε σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2010. Και μετά, λόγω του της Συμφωνίας της Ντοβίλ, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ανταποκρίθηκαν ε, στο πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική περίπτωση. Αυτό έχει τονιστεί από την Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και οι δράσεις μας αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι μια μοναδική περίπτωση. Ακριβώς γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια μείζον επιχείρηση αναδιάρθρωσης του χρέους με μείωση κατά 53,5% που θα μειώσει ε, το χρέος της Ελλάδας, θα κουρέψει το χρέος της Ελλάδας κατά 100 δις ευρώ που είναι η μεγαλύτερη ε, αναδιάρθρωση χρέους στην ε, ιστορία και μια πολύ σημαντική συνεισφορά στη μείωση του βάρους του χρέους που φέρει η Ελλάδα. Ο κ. Γκέμπελς αναφέρθηκε στο θέμα της εξυγίανσης και της ανάπτυξης. Η άποψή μας είναι ότι τα μέτρα εξυγίανσης δεν υποσκάπτουν την ανάπτυξη, την αύξηση της ανάπτυξης και την πρόθεση αυτών των μέτρων. Φυσικά η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση ανταγωνιστικότητας χαμηλή παραγωγικότητα, έχει τεράστιες εξωτερικές ανισορροπίες, καθώς και μια δημοσιονομική κρίση με τρομερά ε, ελλείμματα και χρέη. Η Ελλάδα πρέπει να σημειώσει πρόοδο και στα δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Αυτό είναι σίγουρα εκ των ονουκάνευ. Και το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να εστιάσουμε και στην δημοσιονομική εξυγίανση και σε μέτρα που αυξάνουν την ανάπτυξη. Για να υποστηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, η Κομισιόν δημιούργησε πέρυσι αυτή την ομάδα κρούση, αυτή την task force και αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση επέκταση ε, τη δραστηριότητά τη. Βασιζόμαστε σε... στην πραγματογνωμοσύνη των κρατών μελών της Ευρωζώνης καθώς και στην πραγματογνωμοσύνη του δούνου του ΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών. Και η βασική στόχη είναι καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ίσπραξη εσόδων από τους φόρους, αλλά και για να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη του προγράμματος. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα χρειάζεται, γιατί καταρχάς πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, ούτως ώστε να είναι πιο θετικό για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο ε, πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ο Γιώργα Άσμουσεν, τέσσερα λεπτά. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις. Ο κύριος Γκοζές ρωτά πώς μπορεί να αναπτυχθεί ξανά η Ελλάδα εάν νομίζουμε ότι μπορεί. Εμείς λέμε ναι, σαφώς υπάρχει πιθανότητα το πρόγραμμα να λειτουργήσει. Υπάρχει εγγύηση ότι θα λειτουργήσει, όχι. Το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει εάν εφαρμοστεί 100% σε ολόκληρη την περίοδο και αυτό είναι δυνατόν μόνο εάν σαφώς το δεχτούν το πρόγραμμα σε όλο το ελληνικό πολιτικό φάσμα. Αυτή, η, αν υπάρξει μια πολιτική δέσμευση, αυτή είναι μια διαφορά αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, όπου υπάρχει σαφής πολιτική στήριξη για τις ε, απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις. Αυτό απαιτείται Ε, εάν συμβεί αυτό και είναι ρεαλιστικό το σενάριο για την παγκόσμια οικονομία, που αναμένουμε πως το 2013 θα έχουμε μηδενική ε, ανάπτυξη και θα επιστρέψει η Ελλάδα το 2014 σε θετική ανάπτυξη. Και ρωτάτε τι θα γίνει αν αποτύχει το πρόγραμμα. Εγώ θα προτιμούσα σε μια αρχική βάση του προγράμματος να γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικέ, αυτομάτως η πρώτη μας λύση καταστρέφεται. Τώρα περνάω στις ε, άλλες ερωτήσεις. Ναι, το πρόγραμμα βλέπει μια μεταβολή στην ε, σύνθεση του πώς δημιουργείται η ζήτηση στην Ελλάδα. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ένα έλλειμμα θετικής παραγωγής, δηλαδή βασίζονταν στην κατανάλωση που βασίζονταν με τη σειρά της στην πίστοση και τώρα ε, οδηγεί περισσότερο σε ανάπτυξη που βασίζεται στις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Και με ρωτήσατε εάν εγώ ή εμείς ε, θα συμφωνούσαμε με αυτό το οποίο είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πως χρειάζεται ένα μείγμα ε, και οικονομικής ε, σταθεροποίησης αλλά και όθηση στην ανάπτυξη. Μα πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Αλλά είμαι σίγουρο πως ε, το γνωρίζει αυτό ούτως ή άλλως και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ότι δηλαδή είχε δύο πυλώνες, αυτούς τους δύο πυλώνες, το πρόγραμμα ευθύ εξ αρχής. Και την πτυχή της οικονομίας και την, ε, την ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας για να δημιουργηθεί ανάπτυξη και απασχόληση. Κατόπιν, οι επόμενες ερωτήσεις. Ε, για την αγορά εργασίας και την μείωση τη βραχυπρόθεσμη. Υποθέτω, σύμφωνα με τις προβολές μας, πως το πρόγραμμα θα σταθεροποιήσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας το 2013 και πως η ανεργία μπορεί να αρχίσει να μειώνεται ξανά από το 2014. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η απαραίτητη εξυγίανση βράχει πρόθεσμα είναι αρνητική για την ανάπτυξη. Αυτό το βλέπουμε σε διάφορα προγράμματα προσαρμογής, ανά την Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η εναλλακτική. Εάν η κατάσταση του χρέους είναι μη βιώσιμη, έτσι την κρίνουν οι επενδυτές και οι αγορές, πρέπει να υπάρξει μια εξυγίανση, αλλιώς ποτέ δεν θα ανακτήσεις την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και χωρίς αυτό δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Οπότε πρόθεσμα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη, αλλά μεσοπρόθεσμα θα αποδώσουν οι μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Πολ Τόμσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε για τα όσα έχει κάνει η Τρόικα. Να πω ότι η Τρόικα με τους, ε, είπα, τους ε, αρμόδιους ε, στο Υπουργείο Οικονομικών και με άλλα Υπουργεία που συναντήθηκε. Κυρίως όμως η Τρόικα εργάζεται σε μεγάλο βαθμό παρέχοντας τεχνική συνδρομή και αρρωγή. Ούτε μια εβδομάδα δεν περνάει που να μην έχουμε κάποιου πραγματογνώμονε επαείοντε στην Ελλάδα που να συνεργάζονται με Έλληνε ειδικού και που να εξετάζουν πολύ τεχνικού χαρακτήρα θέματα μέσα από θεσμικά όργανα και θέματα. Και αυτό με οδηγεί σε ένα σημείο επισκοπώντα το τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα. Όλοι συνειδητοποιούμε στην Ελλάδα από πλευρά τη Τρόικα ότι το διοικητικό δυναμικό στην Ελλάδα για την ε, επίτευξη των μεταρρυθμίσεων είναι μικρότερο από αυτό το οποίο αναμέναμε και πρέπει να ανακάμψει η Ελλάδα, η Ελλάδα ώστε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις δράσεις και να υπάρχουν οι ευτές επιπτώσεις. Και αυτό θέλουμε να αντανακλάτε και να επιτευχθεί με το νέο πρόγραμμα. Στο θέμα αυτό φυσικά κατανοούμε ότι η Ελλάδα περνά μια κοινωνικά πολύ οδυνηρή περίοδο και διεργασίες οδυνηρές. Όμως θα πρέπει να το δει κανείς υπό αυτό το πρίσμα. Αυτό συμβαίνει παρόλο το γεγονός ότι η Ελλάδα παίρνει από τους Ευρωπαίους εταίρους, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το, Ευρω... το Ταμείο, πολλά περισσότερα από ό,τι συνήθως δίνονται πραγματικά σε έκτακτη κλίμακα, ξεχωριστή κλίμακα και στα ποσά σε όγκο κεφαλαίων και για τη διάρκεια που προβλέπεται η παροχή τους. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει οδυνηρότατη προσαρμογή. Παρόλες τις προσπάθειες να απαυλύνουμε, να αποσβέσουμε τις, τις επιπτώσεις αυτών των προσαρμογών. Είναι οδυνηρή αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος και να τα καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτυγχάνοντας τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να αποκατασταθεί η οικονομική ανάπτυξη. Έγινε λόγος για τον ελάχιστο μισθό και τους νέους και την καταπολέμηση της ανεργίας. Αυξήθηκε κατά 60% μεταξύ 2000 και 2009 ο μισθός, ενώ είχαμε χαμηλότερο ποσοστό αύξησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελάχιστος μισθός στην Ελλάδα είναι 50% πάνω από τον ελάχιστο μισθό στην Πορτογαλία και δυσανάλογα παραπάνω από, ό,τι στην Ισπανία και 50% πλάσιος ο ελάχιστο μισθό, από ότι ο ελάχιστο μισθό στη Ρουμανία και Βουλγαρία εταίρων στα Βαλκάνια κατανοούμε φυσικά ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο μισθό με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό είναι κλειδί για να μπορέσουν οι επιχειρήσει να απορροφήσουν περισσότερου νέου και να αντιμετωπίσουν έτσι αυτό το οποίο είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση όσον αφορά την ανεργία των νέων σήμερα και απαράδεκτη κατάσταση. Όπως είπα, το πρόγραμμα δεν είναι μόνο η μείωση μισθών. Το πρόγραμμα κυρίως επικεντρώνεται στην διάθεση κονδυλίων σε πιο παραγωγικές χρήσεις, απελευθερώνοντας το μεγάλο δυναμικό της Ελλάδας για να μπορέσει να καλύψει το κενό που την χωρίζει από την ανταγωνιστικότητα και την ε, βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν πιστεύει ότι κάτι λείπει για παιδεία ή τομεί που δεν έχουμε καλύψει και θα έπρεπε να καλυφθούν, εγώ θα σας έλεγα ότι το πρόγραμμα καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων-απαντήσεων. Εδώ θα ακούσουμε έξι ομιλητές, ένα λεπτό καθένας. Θα ξεκινήσουμε από την Επιτροπή την Οικονομική, από την Ομάδα των Φιλελευθέρων, από τον κύριο Σκυλακάκη. Ο, οι κύριοι Άσμουσεν και Τόμσεν μίλησαν για το μεγάλο μέγεθος της κυβέρνησης. Και όμως το 2012 το σύνολο της προσαρμογής στην Ελλάδα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι πρωτογενείς δαπάνες μένουν στο ίδιο επίπεδο, ενώ τα πρωτογενή έσοδα αυξάνονται κατά τρει μονάδες, λόγω νέων φορολογιών, καθώς η φοροδιαφυγή ακόμη δεν αποδίδει. Την ίδια ώρα συνεχίζονται στο δημόσιο τομέα μαζικά οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις σε ηλικίες μέχρι και 52 ετών, με βάση διατάξεις που ψηφίστηκαν υπό την δική σας επίβλεψη της Τρόικα. Επίσης συνεχίζονται και οι προσλήψεις στο δημόσιο. Η δυσανάλογη επιβάρηση του ιδιωτικού τομέα και η μη πληρωμή στο, στον ιδιωτικό τομέα των κρατικών υποχρεώσεων ύψου 3% του ΑΕΠ επιτείνει τη μαζική ανεργία. Καταστρέφονται πλέον δεκάδε χιλιάδε ανταγωνιστικέ θέσει εργασία. Πώ θα προχωρήσουμε για να απορροφήσουμε αυτού του ανέργου, μπορεί να έχει το πρόγραμμα επίδεση επιτυχία χωρί ειδική προσπάθεια για ιδιωτικέ επενδύσει στο πλαίσιο κάποιου είδου σχεδίου Marshall. Και επίση, χθε τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα κατηγόρησαν το ένα το άλλο για 2.500 νέε προσλήψει στα ελληνικά ταχυδρομεία. Ποια είναι η δική σα θέση για τι προεκλογικέ προσλήψει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Από τους Πράσινους, Επιτροπή Απασχόλησης, η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Um, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέρον που ακούσαμε αυτά τα οποία υπόθηκαν για την αύξηση της ε, δυνατότητας ε, τη ελληνική διοίκηση, γιατί ανησυχούμε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και αν υπάρχει ικανότητα απορρόφηση για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτέ τι ευκαιρίε. Πόσο μάλλον ε, που υπάρχουν και οι δυσκολίες χρηματοδότηση, και θα ήθελα κάποια απάντηση. Επίσης, μιλήσατε για ανάπτυξη και δουλειέ. Πώς θα διασφαλίσουμε πώς η ανάπτυξη θα δημιουργήσει δουλειέ. Γιατί μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που δεν θα συνδέεται με αύξηση της απασχόληση. Ποιο είναι υπεύθυνο γι' αυτό και πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτό το θέμα και να υπάρξει ανάπτυξη και να αυξηθούν παραδείγματο χάρη οι ανανεώσιμες για να μειωθούν οι εισαγωγέ ε, καυσίμων. Και μετά για τη φοροδιαφυγή στον ιδιωτικό τομέα, γιατί εάν είναι πραγματικά να δούμε τι γίνεται με τον ιδιωτικό τομέα, σε κάποια άλλα κράτη-μέλη, ε, αν σκεφτούμε τι γίνεται εκεί, δεν τα πάνε και τόσο καλά όσον αφορά την πληρωμή των φόρων. Σας ευχαριστώ για τους... Από την Νομισματική Επιτροπή, από την ομάδα ECR, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ε, για τις τελευταίες ε, προβλέψεις ε, για τα μέτρα για την Ελλάδα με σκοπό την αποκατάσταση. 50 δις προβλέπει το πρόγραμμα για να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν την επίπτωση της ύφεσης και την αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους. Ξέρετε ότι σημαντική είναι, σημαντικός είναι ο δανεισμός των τραπεζών για να υπάρξει νέα οικονομική δραστηριότητα. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι βραχυπρόθεσμα οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή, αλλά είναι και πιο ε, ευάλωτες αν στερεύσει το ρευστό. Επομένως, ε, οι νέοι κανόνες της Βασιλείας 3 για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις και η η εφαρμογή τους ε, θα εξασφαλίσουν αυτό που χρειάζεται. Τι μέτρα ε, προβλέπετε ούτως ώστε ο μελλοντικό δανεισμός των τραπεζών προς τις μικρομεσαίες, επιχειρήσεων, ε, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να, μην, να, να υπάρξει, να είναι διαθέσιμος. Ευχαριστώ από το, τους φιλελεύθερους Επιτροπή Απασχόλησης, η επόμενη ομιλήτρια, Νάτια Χίρς. Κυρία Χίρς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο ήδη προαναφέρθηκε, κυρίως ε, η ανεργία των νέων, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όταν βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει περίπου 50% ποσοστό ανεργία των νέων. Αυτό είναι μια ολόκληρη γενιά που χάνεται. Αν δεν μπορέσει να καταρτιστεί και να εκπαιδευτεί και δεν έχει απασχόληση, περνά το πρόβλημα στα επόμενα 10-20 χρόνια και διαιωνίζεται. Και α το πω έτσι, ακόμα και αν τα άλλα προβλήματα μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όλο και περισσότερο και με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα έχει δραματικές διαστάσεις. Με ενδιαφέρει. Πού βλέπετε δυνατότητες να γίνει κάτι από πλευράς προλαλισσάσης εθέτει ε, το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κυρίως εδώ χρειάζονται υποστήριξη ή δηλαδή και σε άλλο επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ταμεία που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο αλλά με συγχρηματοδότηση πάντα υποχρεωτικά. Κατά πόσο βλέπετε εδώ κάποιε δυνατότητε σε αυτό το θέμα να τύχει αντιμετώπιση και συνέχεια και να μην αφήσουμε μια ολόκληρη γενεά να χαθεί στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ε, Τελευταίος ομιλητής αυτής της ομάδας από τους Πράσινους ε, Επιτροπή, ο Φιλίπ Λαμπέρτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που συνέβη χτες στην Επιτροπή μας. Υπήρχε εδώ πέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ που είπε για την Ελλάδα πως ε, η έλλειψη αναγνώρισης πριν από δύο χρόνια πως είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα και η έλλειψη αναδιάρθρωση του χρέους ήταν το προπατορικό αμάρτημα της Τρόικας στην Ελλάδα και ήταν η μεγαλύτερη ανευθυνότητα των ευρωπαϊκών αρχών και της Τρόικας ε, προς την Ελλάδα. Και όταν σας ακούω σήμερα έχω την αίσθηση πως ε, πάλι τα ίδια έχουμε. Αρνείστε την πραγματικότητα. Εσείς κύριε Άσμουσεν είπατε πως δεν ήσασταν τότε μέλος της ε, ομάδας, αλλά παίξατε ρόλο στην άρνηση αυτή της πραγματικότητας. Και όταν σας ακούω βλέπω ένα πολύ σφιχτό σχέδιο με ε, λίγες ε, δυνατότητες ε, και πιθανότητες όπως λέτε αρνητικών εξέλιξεων. Νομίζω κύριε Τόμψεν είστε πολύ αισιόδοξο τι έχετε προβλέψει ως λύση ανάγκης για τα απρόβλεπτα, όπως παραδείγματο χάρη τη μη εκτέλεση που λέτε πως είναι πρόβλημα ε, στην περίοδο που μας πέρασε και τι σχέδια ανάγκη έχετε σε περίπτωση που αποτύχει το σχέδιο σα. Πράγματι, καλά λέτε κυρία Άσμουσεν, δεν πρέπει να εξετάζουμε εναλλακτικέ ΒΓΔ, αλλά επειδή και το δικό σα το ιστορικό όσον αφορά τι προβλέψει σα δεν είναι τόσο καλό, δεν σα εμπιστευόμαστε και τόσο. Λοιπόν, θα απαντήσουν σε αυτέ τι πέντε ερωτήσει καταρχήν όλοι Ρεν. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την ερώτηση της κυρίας Σουινμπέρν για την ακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και μετά θα περάσω στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Η οικονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική σταθερότητα ήταν βασικό στοιχείο, βασικό στόχος του προγράμματος. Μόνο σε ένα περιβάλλον χρηματοπιστωτικής σταθερότητας οι τράπεζες μπορούν να παίξουν το ρόλο τους που είναι να δώσουν πίστοση στην πραγματική οικονομία και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Από την αρχή του προγράμματος, τα εξαιρετικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από την ΕΚΤ έχουν εξασφαλίσει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε αρκετή ρευστότητα και παρότι το πρώτο πρόγραμμα έχει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό δεν άρκεσε και αυξήθηκε στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο σημερινό πρόγραμμα. Κάτω την άποψή μα, αυτό είναι επαρκέ για να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζε έχουν ε, είναι παρκώ ανακεφαλαιοποιημένε για να αντιμετωπίσουν την ύφεση, να αντιμετωπίσουν τα επισφαλή δάνεια και τι απώλειε λόγω τη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, Βάσει των διαρθρωτικών ταμείων δημιουργήθηκε ένα νέο ταμείο εγγύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το νέο μέσο θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση αρκετά έντονα να έχουν πρόσβαση σε πίστη χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα για το ελληνικό κράτος και ευθύνε για το ελληνικό κράτος. Μέχρι το 2015 η συνολική πίστη που θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα φτάσει στο 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα της συγχρηματοδότησης και των διαρθωτικών ταμείων. Να σας ενημερώσω ότι μετά την πρωτοβουλία του Ιωάννης Χάρν, διάφορα προγράμματα 181 προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό αποφασίστηκε και το ύψος των κονδυλίων είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν για αυτά τα προγράμματα. Ο ε, σκοπός είναι να δοθεί νέα όθηση ε, στην ε, υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαφορετικά ταμεία. Μιλάμε για προγράμματα που θα έχουν σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αυτό συμπεριλαμβάνει τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, καθώς και ο τουρισμός ε, και κοινωνικά προγράμματα επίσης. Δεν υπάρχουν νέα έργα και αυτό βοηθάει γιατί έχει προχωρήσει αρκετά ο σχεδιασμός και απλώς ε, περιμένουμε τώρα να μπούμε στη φάση της εφαρμογής. Μιλάμε για σχέδια και προγράμματα τα οποία θα προωθηθούν, ε, που επιλέγησαν από χιλιάδες. Και αυτά θα απορροφήσουν περίπου το μισό διαθέσιμο χρήμα. Οι ελληνικές αρχές ε, παρακολουθούν το θέμα και την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων εκ του σύνηγης με την υποστήριξη των υπηρεσιών της ε, Κομισιόν. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης, μια πρώτη έκθεση αυτή τη στιγμή την οριστικοποιούν οι ελληνικές αρχές και θα τη λάβετε σύντομα. Από ό,τι φαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή εξυπηρετεί ακριβώς το στόχο με αποτελεσματικότητα, δηλαδή εστιάζει σε πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες, ούτως ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση. Ευχαριστώ. Τέσσερα λεπτά και ο κύριος Άσμουσεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα της απασχόλησης στο δημόσιο. Η γεγονός είναι πως ε, στο πρώτο πρόγραμμα η μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο δεν ήταν αυτή η οποία είχε αναλυφθεί ως δέσμευση και τώρα προσπαθούμε με το δεύτερο πρόγραμμα να διορθώσουμε την κατάσταση έτσι ώστε να γίνει προσαρμογή και στον δημόσιο τομέα. Αυτό είναι απαραίτητο. Σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους, το μέγεθος του ελληνικού δημοσίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλήσατε για τις προεκλογικές προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Για να είμαι ειλικρινής δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω. Ζητήσατε ένα σχέδιο Μάρσαλ, ένα είδο σχεδίου Μάρσαλ. Συμφωνώ πω υπάρχει ανάγκη επενδύσεων, αλλά θέλω να είμαι σαφή για ε, δημόσιες επενδύσεις δεν προβλέπονται, επιπλέον δημόσιες επενδύσεις δεν προβλέπονται λεφτά στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει χάσει πρόσβαση ε, στις αγορές και βασίζεται για μια χρηματοδότηση εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα στους εταίρους της και στο δυνατό. του. Οπότε, οποιοδήποτε αίτημα για περαιτέρω χρηματοδότηση σημαίνει περισσότερα λεφτά από τους Ευρωπαίους εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οπότε, δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό. Για τα κονδύλια, τα κοινοτικά, το κάλυψε ο Επίτροπος. Το θέμα είναι, ναι, πρέπει να φροντίσουμε ε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, να δημιουργούν ε, δουλειά και στο πρόγραμμα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα διαφορετικών μεταρρυθμίσεων που προωθούν την απασχόληση, μεταξύ των οποίων ένα πρόγραμμα Fast Track για νέα έργα, η δημιουργία μίας θηρίδας για την δημιουργία νέας εταιρείας και για τις εξαγωγές και ε, προγράμματα για να ανοίξουν διάφορες αγορές όπως κλειστά επαγγέλματα όπως οι αρχιτέκτονες κτλ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως προϋπόθεση για να δοθεί πίστοση στην ελληνική οικονομία και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα από είναι ένας από τους γρήγορους στόχους που έχουμε θέσει στο δεύτερο πρόγραμμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ε, που επιβλέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα δει μέχρι το τέλος Μαρτίου ποιες τράπεζες είναι βιώσιμες και ποιες όχι. Αυτές που θεωρούνται βιώσιμες αμέσως θα ανακεφαλαιοποιηθούν ή δυνατόν μέσω των ιδιωτικών αγορών, εάν όχι ε, μέσω κονδυλίων του προγράμματος, ήδη μέσω της πρώτης δόσης, για να διασφαλιστεί πως ε, έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση, μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο τους, να δανείσουν στην πραγματική οικονομία και να είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε, ε, στις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν ήδη λοιπόν από την πρώτη δόση διαθέσιμα κονδύλια. Η δεύτερη δόση η οποία θα εκταμιευθεί μετά την πρώτη εξέταση του προγράμματος. Έχει πάλι το ίδιο ποσό, 25 δισεκατομμύρια χοντρικά, για την ανακεφαλαιοποίηση των ε, τραπεζών και όλα αυτά το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ένας τομέας δηλαδή όπου θα κινηθούμε γρήγορα με το νέο πρόγραμμα. Ο κύριος Λάμπερτς ρώτησε, δήλωσε μάλλον, πως αρνούμαστε την πραγματικότητα. Δεν είμαι σίγουρος. Και άλλοι άνθρωποι έχουν πει πως αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. Εάν δείτε τι έγινε σε άλλα προγράμματα στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία, η δήλωση αυτή είναι πάρα πολύ σπάνια. Οπότε, ναι, το πρόγραμμα κινδυνεύει από προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά θεωρούμε πως είναι βιώσιμο, θα είναι βιώσιμο το χρέος το 2020 εάν εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα. Οπότε δεν βλέπω έλλειψη ρεαλισμού υπονοήσατε κάτι για την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό βασίζονταν κυρίως σε ανησυχίες για μετάδοση του προβλήματος σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Νομίζω λοιπόν ότι με το τείχος προστασίας που δημιουργήσαμε περιορίσαμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε μετά να αντιμετωπίσουμε το μη βιώσιμο χρέος της Ελλάδας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Τόμσεν τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε μόνο μία σύντομη προσθήκη σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα όσον αφορά τις πιστώσεις ε, για τις επιχειρήσεις ε, και τις τράπεζες. Ένα από τα πράγματα που είναι καινούριο σε αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη, σε αυτή τη συγκυρία, είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διεθνώς επαΐοντες ε, που θα εξετάσουν τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων. Ένα από τα προβλήματα, και αυτό είναι μια τάση τραπεζών, να έχουν διάβλους που θα δίνονται, να υπάρχουν δάνεια και πιστώσεις που θα δίνονται στις ε, ε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πρέπει όμως ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα των μη βιώσιμων επιχειρήσεων ε, και το θέμα της δανειοδότησής, μου, δανειοδότησής τους. Εξετάζοντας τα λογιστικά αυτών των ε, ε, τραπεζών και επιχειρήσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η πτυχή. Θα ενθαρρυνθούν τράπεζες στο μέλλον να διοχετεύουν πιστώσεις σε πιο δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η καλύτερη μελλοντική προοπτική. Να υπάρχουν αυτές οι διατάξεις ε, και οι ρήτρες ώστε όταν θα δίνεται πίστοση σε μία μη ανταγωνιστική επιχείρηση απαιτεί εγγυήσεις και έτσι γίνεται πιο ακριβή η δανειοδότηση πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ρήτρε και ασφάλειε που θα ε, λειτουργήσουν μέσω αυτού του προγράμματο ώστε να διοχετεύονται μέσω διάβλων τα δάνεια επιστώσει αυτέ σε δυναμικέ μικρομεσαίε επιχειρήσει ώστε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Τώρα, θα ήθελα για το επόμενο θέμα να σα καλέσω να κοιτάξετε, την, να διαβάσετε την έκθεσή μα. Έχει ένα μεγάλο παράρτημα. Δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών αναφέθηκε. Και αυτό είναι μάλλον ε, κάποια κατεφημισμών διατύπωση. Θα δείτε ότι η κύρια ευαισθησία εδώ είναι το θέμα των διαθωτικών μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Οποιαδήποτε αποτυχία να αναζωογονηθούν οι μεταρρυθμίσεις, οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι κύρια προϋπόθεση του νέου προγράμματος πραγματικά θα κάνει μη βιώσιμο το χρέος και πολύ γοργά κιόλα μάλιστα. Τώρα, τι θα συμβεί και τι συμβαίνει αν η Ελλάδα κάνει τις καλύτερες προσπάθειες από πλευράς της, όμως υπάρχουν αντίξωες συγκυρίες και αντίθετοι άνεμοι και θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν και είπαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ελλάδα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές υπό την προϋπόθεση και υπόθεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις από πλευρά τη. Πλήρω. Αυτό είναι το, η, το στοιχείο που έχει σημασία κλειδιού και η ρήτρα ασφάλεια. Εφόσον κάνει η Ελλάδα αυτό το οποίο χρειάζεται και πρέπει να κάνει, η Ευρώπη θα την υποστηρίξει. Και αυτό είναι το, η ακρογωνία λίθο όσον αφορά την ε, συνέχιση αυτή τη προσπάθεια. Οι Έλληνε είναι υπεύθυνοι να το κάνουν. Ευχαριστώ. Um, Πιέζει ο χρόνος και περνάμε τώρα στον τρίτο γύρο ερωτήσεων. Και πάλι τώρα θα έχουμε ένα λεπτό ανά τέσσερις αγορητές και θα δώσουμε στους ε, όσοι μετέχουν εκπροσώπους ε, τρία λεπτά στον καθένα να απαντήσουν. Ο, ο Νίκλας είναι ο πρώτος, θα έχει δύο ερωτήσεις, δύο λεπτά θα έχει λοιπόν για να τις διατυπώσει. Έχει τον λόγο Νίκλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριος Χουντής παρακαλώ, Νίκος Χουντής. Έχω μαζί μου την πιο διάσημη φωτογραφία που κυκλοφορεί για σας στην Ελλάδα. Είναι τότε που με διαγράμματα και πίνακες λέγατε ότι με βάση το πρόγραμμα της Τρόικα η ύφεση θα σταματήσει το 2011 και ότι το 2012 θα έχουμε ανάπτυξη 1,2. Αυτά λένε τα διαγράμματά σας, αυτό δείχνει η φωτογραφία σας. Φυσικά αντί για ύφεση, ανάπτυξη έχουμε ύφεση. Η ύφεση έχει φτάσει στο 7%. Έχουν κλείσει χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις. Υπάρχουν πάνω από 20% άνεργοι και άνεργοι νέοι. Χιλιάδες άστεγοι και άποροι. Ένας λαός δυστυχισμένος και προσοδευμένος. Έχετε αποτύχει ικτρά. Τα περί δεν ισχύουν διότι θα έρθει η ώρα και θα κουβεντιάσουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, επομένως δεν είναι σοβαρή επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά επιμένετε. Με βάση λοιπόν το νέο μνημόνιο προβλέπεται περικοπή 12 δις για το επόμενο διάστημα που σημαίνει μειώσεις πάλι συντάξεων, ε, απολύσεις στο δημόσιο, μειώσεις κοινωνικών δαπανών που σημαίνει και άλλα χρήματα θα φύγουν από την ελληνική οικονομία και θα μπει ή θα συνεχίσει να λειτουργεί ο φαύλος κύκλος της ύφεση και του δανεισμού και των ελλημάτων για την Ελλάδα. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω και που είναι όχι δικό μου, όλο του ελληνικού λαού. Οι μισθοί έχουν μειωθεί. Κατά 22% έχετε καταργήσει τις συλλογικέ συμβάσεις, θέλετε να τους μειώσετε ακόμα περισσότερο. Το είπε ο κύριος Τόμσεν σήμερα, το λέει η έκθεση της Κομισιόν, συγκρίνεται τους μισθούς της Ελλάδας με μισθούς άλλων χωρών όπως τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Τι σύγκριση είναι αυτή. Αν βάλετε ένα πρωτοετή θα σας πει είσαστε είσαστε από το μάθημα. Και μπαίνω στο ερώτημά μου, διότι δεν με απασχολεί αυτό. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν είναι στόχος της Τρόικα όπως πιστεύει ο ελληνικός λαός ότι θέλετε να πάτε τους μισθούς στην Ελλάδα στο επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που είναι 150 ευρώ το μήνα ότι δεν θα πάτε τις εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες νοτιοανατολικής Ασίας. Thank you. Στο. Περιμένω την ε, διερμηνία μου να τελειώσει. Από την EFT, την κυρία Νίκη Τσαβέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Για ποια ελληνική ανταγωνιστικότητα μιλάμε. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε δηλώσεις σχεδόν απειλητικές, σχεδόν εκβιαστικές από Ευρωπαίους αξιωματούχους από το Συμβούλιο για την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ. Οι δηλώσεις αυτές έπληξαν κέρια το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας και των Ελλήνων διεθνώς, επιτείνοντας το οικονομικό μας πρόβλημα Ποιος επενδυτής θα επενδύσει σε μια χώρα που επίκειται να βγει από το ευρώ. Κάποιοι λοιπόν από το Συμβούλιο, το τονίζω, κατέστρεψαν τον ευρωπαϊσμό, την αξιοπρέπεια και το αίσθημα ασφάλειας του ελληνικού λαού πράγμα το οποίο θα το δούμε στις επικείμενες εκλογές. Από χθε όμως έχουμε δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε, του κυρίου Γιούνκερ ότι ποτέ το σενάριο για έξοδο από το ευρώ δεν ήταν ρεαλιστικό. Ποιο λοιπόν ισχύει, μπορείτε να μας πείτε, είναι ρεαλιστικό το σενάριο της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ ή όχι. Ευχαριστώ. Thank uh, and ομιλητής αυτό από την e Έχουμε μεγάλη οικονομική κρίση την οποία δημιουργήσαμε μόνοι μας. Ε, είμαστε στο δέκατο ο έτος ενός καταστροφικού πειράματος με ένα νόμισμα το οποίο οποιοδήποτε μαθητής έβλεπε πως θα αποτύχανε. Ένα πολιτικό επιχείρημα επικίνδυνο όπως απέδειξε η του 1920 και του 30. Και τι κάνουμε εδώ πέρα, επιδοτούμε τράπεζες και κεντρικές τράπεζες με τα λεφτά των φορολογουμένων, αυτοκτονίες, εγκαταλείψεις παιδιών, 50% ε, αύξηση της ε, ανεργίας των νέων ε, στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει εάν η Ελλάδα είναι μοναδική. Δεν νομίζω να είναι μοναδική. Είναι απλά το πρόβλημα το τρέχον δεν βλέπει το Διεθνή Νομισματικό Ταμείο πω το σύστημα έχει αποτύχει και θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι χρεοκοπημένε οικονομίε να ξαναρχίσουν με το δικό του νόμισμα και ερετού δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτε. Θα περάσουμε τώρα στι απαντήσει, ξεκινώντα από την ε, Κομισιόν μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τέλο το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Όλοι. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα για το ερώτημα του κ. Χουντή για τις προβλέψεις της ανάπτυξης. Είναι γεγονός πως οι προβολές ε, ανάπτυξης ε, της ε, Τρόικας του Μαΐου του 2010 ήταν υπερβολικά αισιόδοξε. Πολλοί παράγοντες συνετέλεσαν σε αυτό. Στο να είναι δηλαδή το αποτέλεσμα χειρότερο από ό,τι είχαμε αρχικά προβλέψει. Ένας παράγον ήταν η συζήτηση εμπλοκής ε, του δημοσίου τομέα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή που ενίσχυσε την οικονομική αβεβαιότητα και απέφευγαν να αναλάβουν κίνδυνο οι επενδυτές και οι καταναλωτές όπως ε, θυμόμαστε ε, από τον καιρό του Οκτωβρίου 2010 της Συμφωνίας της Ντοβίλ κάτι το οποίο ενισχύθηκε από την έλλειψη ευρείας ε, συνένεσης ε, για πολλές μεταρρυθμίσεις κλειδιά που ήταν στο πρώτο πρόγραμμα. Και βεβαίως υπήρχε και η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα που έπαιξε ένα ρόλο. Ως αποτέλεσμα δεν σημειώθηκε επαρκής πρόοδος ε, σε πολλές ε, μεταρρυθμίσεις ε, διαρθρωτικές οι οποίες θα ενίσχυαν την ανάπτυξη, κάτι το οποίο επιδεινώθηκε και από την ε, χαμηλή διοικητική ικανότητα στην εφαρμογή τους. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχική μου παρέμβαση, υπάρχουν, υπήρχαν δύο αχίλιες φτέρνες. Η μία είναι η έλλειψη πολιτικής ενότητας και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο οι Έλληνες, οι Έλληνες πολίτες και ολόκληρη κοινωνία μπορεί να διορθώσει γιατί αυτό απαιτείται για να υπάρξει στήριξη για ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα οικονομικής ε, μεταρρύθμισης και προσαρμογής. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε την ασθενή διοικητική ικανότητα της Ελλάδας, κάτι το οποίο κάνουμε με την ομάδα δράσης ε, στην Ελλάδα που στόχο έχει να στηρίξει την Ελλάδα στους στόχους αυτούς. Δεύτερον, για τους μισθούς ε, και την ανταγωνιστικότητα. Ενώ οι μεταρρυθμίσεις του πρώτου προγράμματος βοήθησαν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα ως ένα βαθμό, το υπόλοιπο κενό της ε, ανταγωνιστικότητας ε, υφίσταται και μετριέται στο μοναδιαίο κόστο εργασία. Το να κλείσει αυτό το κενό εντός τη Ευρωζώνης ε, θα απαιτήσει μια ακόμη πιο έντονη εσωτερική υποτίμηση από την Ελλάδα και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δεύτερου προγράμματος. Η συμφωνημένη προσαρμογή των μισθών ε, στον ιδιωτικό τομέα και η τροποποίηση των ε, διαδικασιών ε, καθορισμού του μισθού συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων και διατησίας αποτελούν βασικά στοιχεία της προσπάθειας επιτάχυνσης της εσωτερικής υποτίμησης. Όμως η μείωση του κόστους ε, του μισθολογικού δεν θα μπορέσει να προωθήσει την ανάπτυξη και τις δουλειές αν δεν συμπληρωθεί από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες και τις αγορές για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και η παραγωγικότητα. Και αυτά αποτελούν μέρος του δευτέρου προγράμματος. Όπως ε, είπαν και οι κύριοι Άσμουσεν και Τόμσεν, το δεύτερο πρόγραμμα έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο ως προς την εφαρμογή του. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενισχυμένη πολιτική ενότητα στην Ελλάδα και με συνεχή αποφασιστικότητα για να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα της χώρας. Έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να μεταρρυθμιστεί και να συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Και τώρα ο επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ. Μπορεί να είμαι σύντομο, γιατί προσυπογράφω απόλυτα αυτά που είπε ο Λιρέν. Το πρώτο πρόγραμμα δεν είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, γιατί κυρίως υπήρχε ελληματική εφαρμογή. Το πρόγραμμα προσαρμογής δεν είναι αυτό που δημιουργεί την μείωση και τη συρρήκνωση του ΕΠ. δείχνει απλώς την σοβαρότητα των μακροοικονομικών ανισορροπιών που έχουν σωρευτεί επί σειρά ετών στην Ελλάδα. Και αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί μόνο σε λίγους μήνες. Έτσι λοιπόν ε, οι στόχοι ανάπτυξης του πρώτου προγράμματος όντως δεν επιτεύχθησαν, αλλά λόγω έλλειψης εφαρμογής. Θέλω να είμαι πολύ σαφής, παρότι έχουμε κάποιες διαφωνίες μεταξύ μας. Το PSI έγινε στην Ελλάδα με, και είναι μια μοναδική προσπάθεια, ένα μοναδικό πείραμα. Δεν έχουμε σκοπό να το ξανακάνουμε. Το λέω ξεκάθαρα. Ήταν μια μοναδική απόπειρα, ένα μοναδικό πείραμα και δεν έχουμε σκοπό να το επαναλάβουμε. Ακούστηκε μια ερώτηση ε, ειδικού ενδιαφέροντος για την ΕΚΤ, για την Ελλάδα και την πιθανότητα να φύγει από το ευρώ. Είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση ότι έχουμε το σαφή σκοπό να κρατήσουμε την Ελλάδα εντός του ευρώ, εντός της ευρωζώνης και αν αυτός είναι ο σκοπό μας, τελικά απόκειται στι ελληνικές αρχές και στον ελληνικό λαό να το αποφασίσουν. Ε, υπάρχει ένας ε, τρόπος να παραμείνουν εντός του ευρώ. Το συζητήσαμε. Η περαιτέρω εσωτερική υποτίμηση. Αυτό ε, έχει να κάνει με το κόστος το μισθολογικό, το κόστος των μισθών. Είναι ο μόνος τρόπος ε, με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας μαζί με άλλες μεταρρυθμίσεις ε, που ανέφερε ο Τόμσον στην πρώτη παρέμβαση, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος εργασίας, υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε να κάνουμε όμως μια ουσιαστική εσωτερική υποτίμηση, ούτως ώστε να ανακτήσει η Ελλάδα την ανταγωνιστικότητα εντός της ζώνης του ευρώ. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Γι' αυτό το είπα δύο φορές στην παρέμβασή μου, ότι θέλουμε μια λύση εντός της ευρωζώνης. Γιατί αν μια χώρα από την ευρωζώνη αυτό θα έχει άπειρους κινδύνους ό,τι αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη Ευρωζώνης συνολικά. Και εγώ συστήνω πραγματικό, πραγματικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε έτσι ελαφρά την καρδία για αυτό το θέμα. Είτε μιλάμε για συντεταγμένη χρεοκοπία, είτε για οτιδήποτε. Εάν φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, ε, η χρεοκοπία θα είναι πάρα πολύ άτακτη και πολύ προβληματική. Και γι' αυτό το πρόγραμμα έχει το βασικό στόχο να κρατήσει την Ελλάδα εντό τη Ευρωζώνη, ούτω ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη εν γέννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε κυρία Άσμουσεν, επειδή γνωρίζουμε ότι τώρα θα πρέπει να φύγετε για να μπορέσετε να ε, ταξιδέψετε. Τώρα έχει τον λόγο ο κύριος Πορτόνσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ελληνικό πρόγραμμα αφορά τον εξυγχρονισμό της οικονομίας για βαθύτατες μεταρρυθμίσεις διαδοτικές. και δεν είδα κανέναν πολιτικό, δεν συνάντησα κανέναν υπεύθυνο πολιτικά που θα πιστεύε ότι η εγκατάλειψη της Ευρωζώνης θα διευκολύνει τέτοιες μεταρρυθμίσεις και θα ανακουφίσει. Η Ελλάδα χρειάζεται, πρέπει να εξυγχρονιστεί για να μπορέσει να ανταγωνιστεί στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Τώρα, τώρα για το θέμα του γιατί το ΑΕΠ συνέχισε να μειώνεται παρόλες τις προσδοκίες από το προηγούμενο πρόγραμμα που είχαμε. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό, έχει δίκιο ο κύριος Άσμουσεν σε σχέση με το πρόγραμμα. Αφορά την μη υλοποίηση των μέτρων στη διαθροτική πλευρά των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Έκανε πολλά για την δημοσιονομική εξυγίανση η Ελλάδα, όμως στις μεταρρυθμίσεις χόλενε. Εδώ λοιπόν, ενώ πιστεύαμε ότι οι μεταρρυθμίσει θα είχαν φτάσει σε μια κρίσιμη μάζα και θα υπήρχε βελτίωση και θα υπήρχε σταδιακή αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών. Λόγω τη έλλειψη αυτή τη κριτικής κρίσιμης μάζας υπήρξε αυτή η φθήνουσα πορεία και η συρρήκνωση του ΑΕΠ. Τώρα, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το νέο πρόγραμμα θα πετύχει μόνο αν αναχαιτήσουμε αυτή την εξέλιξη και έχουμε μια αναζωγόνηση διαθωτικών μεταρρυθμίσεων. Ουσιαστικά έχει ένα χάσμα μεταξύ του μισθολογικού κόστου των μισθών και τη παραγωγικότητα η Ελλάδα. Η ακραία επιλογή είναι ή θα είναι πιο παραγωγική η Ελλάδα ή θα μειωθούν αμέσω οι μισθοί. Θα πρέπει να διευκολύνουμε να γίνει η Ελλάδα πιο παραγωγική. Συμφωνούμε όλοι ότι υπήρξαν πολλέ ε, προσαρμογέ ε, με μια υφεσιακή εξέλιξη, με χαμηλού μισθού, μείωση των μισθών το πρόγραμμα όμως στοχεύει στο να αναχαιτιστεί αυτή η εξέλιξη, δημιουργώντας έστω και με καθυστέρηση όλα εκείνα τα μέτρα που θα υλοποιηθούν ώστε να υπάρξει σε ευρύτατο φάσμα ανάκαμψη όσον αφορά τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά βρίσκονται σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει όμως πανάκια, δεν υπάρχει ε, ε, συντόμευση, σύντμηση του δρόμου και μαγική ράβδος. Πρέπει όλα αυτά τα μέτρα στο εύρος τους ε, να υλοποιηθούν. Αν εξετάσετε το πρόγραμμα προσεκτικά, αυτά εμπεριέχονται εκεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Περνάμε στον τελευταίο γύρο τώρα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιες διαδικασίες, κάποιες παρεμβάσεις με το catch the eye που θα δει η πρόεδρος ποιοι ζητούν. Είδαμε τώρα, δεν χρειάζεται να επιμείνετε. Ένα λεπτό για το ΕΛΚ για την απασχόληση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πουπάκης παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ε, θα ρωτήσω κατευθείαν. Πώς αξιολογείτε εσείς τις κοινωνικές επιπτώσεις της συνταγής των μέτρων που επιβάλλετε. 21% ανεργία, ένας στους δύο νέους άνεργος να μεταναστεύει. Άστεγοι, συσίτια, αφού το 30% των συμπολιτών μας, και αυτό δεν το είπατε, είναι κάτω από τα όρια της φτώχεια. Τι άλλο εσωτερική υποτίμηση σήμερα αναφέρεται. Όταν λέτε ότι είμαστε στα μισά της διαδρομής, όταν η χώρα βουλιάει στην ύφεση, το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάζουν λουκέτο στο τέλος του χρόνου, συνεχείς φόροι, καθημερινά χαράτσια που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Πώ είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ενώ διακηρύσει κοινωνικό διάλογο εν τούτης, να καταργεί ομόφωνε κοινωνικέ συμφωνίε και, κοινωνι... και συλλογικέ συμβάσει. Τέλο, πιστεύω ότι δεν μπορεί να αφήνεται από κανέναν ένα λαό να υποφέρει για να ικανοποιούνται οι υπολογισμοί ορισμένων οικονομολόγων και να μην λαμβάνεται υπόψη ότι πίσω από του αριθμού κρύβονται ανθρώπινε ζωέ που τα περιθώρια ανοχή και αντοχή του έχουν εξαντληθεί, ενώ οι πολίτες οδηγούνται στην εξαθλίωση, δεν βλέπουν φως στο τούνελ παρά τις σκληρέ θυσίε που τους επιβάλλονται. Βεβαίω και υπάρχει αναγκαιότητα δημοσιονομικής προσαρμογή. Ο στόχο όμως αυτός είναι εφικτό μόνο μέσα από την υιοθέτηση ενός νέου μείγματος αναπτυξιακής πολιτικής και διαφύλαξης τη κοινωνική συνοχή. Σα ευχαριστώ. Thank you. Uh, now for the Από σοσιαλιστές, η Ελίζα Φερέιρα, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι... Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι μείωσε το έλλειμμα τη ε, κατά 4,2% μέσα σε δύο χρόνια η Ελλάδα έκανε μια διοικητική μεταρρύθμιση μοναδική και ξεχωριστή. Και αυτές οι μεταρρυθμίσει δείχνουν ότι η Ελλάδα έκανε περισσότερα από ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και δεν υπάρχει ισότιμο ε, συγκρίσιμο στοιχείο από άλλες χώρες. Και γι' αυτό ερωτώ, γιατί η Τρόικα δεν το ομολογεί και δεν παραδέχεται ότι σε όρους ανάπτυξης οι δικές της προβλέψεις είναι διαρκώς λανθασμένες. Όταν είναι λανθασμένες οι προβλέψεις λέτε ότι φταίνε εκείνοι που δεν υλοποίησαν. Όμως η Ελλάδα υλοποίησε αυτά τα μέτρα και όσο περισσότερο υλοποιεί η Ελλάδα χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα υπό αυτούς τους όρους σε μια χώρα που εξάγει 20% αυτών που παράγει. Πώς μπορεί να προβλεφτεί μια αύξηση που ο κινητήρας αυτής της αύξησης είναι οι εξαγωγές Μήπως μπορεί να παραδεχθεί καμιά φορά η Τρόικα ότι έκανε λάθος. Μήπως βλέπει η Τρόικα την αξιοπιστία των απαντήσεων που δίνονται όσον αφορά τους εκπροσώπους της Ευρώπης για μια χώρα που είναι μέλος ε, της ζώνης ευρώ. Ευχαριστώ. Το Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, έχουμε ήδη κάνει μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια θέματα. Σύμφωνα ε, με, το δεύτερο πρόγραμμα της οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Τόμψεν ιδιαίτερα, είναι η πρώτη φορά που η επαναδιαπραγμάτευση της νομοσυνομικής στρατηγικής δεν συνοδεύτηκε από αύξηση φόρων, τονίζοντας δε ότι το περιθώριο επιβολής υψηλότερων φόρων και οριζόντιων περικοπών έχει εξαντληθεί. Συμπληρώνεται δε ότι ε, το δημοσιονομικό ελληνικό πρόγραμμα από την αρχή είχε προβλέψει προσαρμογή με κύρια κατεύθυνση την περικοπή δαπανών. Εδώ διαπιστώνουμε, θα το πω και εγώ ακόμη μια φορά, μια στρέβλωση. Πού οφείλεται, πού είναι οι ευθύνε. Κάναμε την αυτοκριτική μα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πού οφείλεται αυτή η στρέβλωση στην εφαρμογή της δημοσιονομική ε, ε, προσαρμογή, στην έλλειψη ε, ε, μεταρρυθμίσεων ε, αναπτυξιακών μέτρων παράλληλα στις μη καλές προβλέψεις για το κόστος το οικονομικό και το κοινωνικό. Τα συμπεράσματα που εξάγονται ήθελα να δω και επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε εν ώψη των νέων μέτρων και περικοπών των δαπανών στο νέο πρόγραμμα τι έχει προβλεφθεί για την προστασία των επενδύσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας για να... και όχι όπως είπε Please don't you lose your discipline at the end. Χάνετε τώρα στο τέλος την ε, πειθαρχία σας, θέλουν και άλλοι να μιλήσουν. Θα ακούσουμε δύο ακόμα μιλητέ γιατί είχαμε τόσους ε, Έλληνες συναδέλφους που μίλησαν. Η Άννη Ποδηματά. One minute. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι ε, ακόμα πιο σύντομη. Το θέμα είναι για όλους το ζητούμενο να εξασφαλιστούν οι προποθέσει επιτυχίας του προγράμματος, αυτού του δεύτερου προγράμματος που συζητάμε, ώστε οι θυσίε των ανθρώπων να πιάσουν τόπο. Και το κλειδί γι' αυτό είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων και των πολιτικών που συμφωνούμε, ε, όπως επίσης και η κοινωνική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που συμφωνούμε, διότι αυτά τα δύο είναι προϋπόθεση για να υπάρχει κοινωνική αποδοχή, αίσθημα ιδιοκτησίας του προγράμματος, που υπογραμμίστηκε και από τους τρεις σας στις παρεμβάσεις σας πριν. Ας αφήσουμε ε, τις ευθύνες στο εθνικό επίπεδο καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών. Θέλω να σας ρωτήσω, τι μπορούσε να γίνει από την δική σας πλευρά και τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τα μέτρα, τι μπορείτε εσείς να κάνετε για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της φοροδιαφυγής και για έναν πιο δίκαιο επιμερισμό του κόστους που είναι προϋπόθεση για να υπάρξει αποδοχή του προγράμματος από την κοινωνία. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ακόμα μιλητές. Παρακαλώ σύντομη να είστε. Χατζημαρκάκη, Κοστέλο και ο Λίαμ κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Τόμψεν που παραδέχτηκε, παραδέχτηκε στο βήμα πριν από λίγες ημέρες πως η Τρόικα έκανε κάποια λάθη. Ένα από αυτά τα λάθη ήταν πως ε, σκέφτηκε πως η ελληνική διοίκηση είχε την ικανότητα να κάνει, να επιτελέσει αυτό το έργο. Και λέτε πως ε, θα, αν τα ξανακάνατε, θα κάνετε τα πράγματα διαφορετικά. Μα θα μπορούσατε να το ξέρετε γιατί ο ΣΑ έβγαλε μια έκθεση πρόσφατα πως 95% της ελληνικής διοίκησης είναι λίγο πολύ άχρηστη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Άλλαξε αυτό τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Έχετε σχέδια να στείλετε Έλληνες από το Δούνου του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσουν την ελληνική διοίκηση το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω, είμαι Ιρλανδέζα ε, μια χώρα δηλαδή του προγράμματος και παρά το ότι δεχόμαστε πως ε, απαιτείται δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να πω πως ε, η οικονομική θέση πολλών χωρών είναι αποτέλεσμα της κρίσης όχι αιτία της. Παραδείγματο χάρη πριν από την κρίση ο λόγος ΑΕΠ προς χρέος Ιρλανδίας ήταν 25% και συμφωνούμε πράγματι πως πρέπει να υπάρξει μια αναπτυξιακή στρατηγική και έχω άρα κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να μας πείτε ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε να λάβετε για την ανεργία των νέων και αν υπάρχουν νέα μέτρα, νέα κονδύλια ή απλά τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Κατόπιν, ε, έκθεση Κορνίλσεν 15 Φεβρουαρίου, την οποία ψηφίσαμε, ε, λέει πως θα πρέπει να εμπλακεί το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Τι άποψη έχει η Τρόικα. Κατόπιν, τι άποψη έχετε για τη δημοκρατική λογοδοσία ως ε, βουλευτής από μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα αυτά νιώθουμε και πονάμε πάρα πολύ για την απώλεια της ε, κυριαρχίας μας και η στάση του Δούνου του, Δούνου του και η νοοτροπία της ε, το επιτείνει ακόμα αυτό. Σας ευχαριστώ όλοι. Ευχαριστώ Σάρον. Αγαπητοί κύριοι, η πολιτική των ε, μεταρρυθμίσεων που συστήνεται λειτουργούν υπό κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς η μείωση των μισθών να κατανέμεται ε, μεταξύ ε, μείωσης των τιμών και αύξηση των κερδών, οι επενδύσεις να είναι ουσιαστικοί και να επωφεληθεί από τη μείωση των μισθών και στην αύξηση των κερδών και οι εξαγωγές να προωθηθούν αν υπάρχει εξωτερική ζήτηση. Ε, αν σκεφτώ ε, αυτά τα τρία σημεία. Ε, το πρώτο δεν ισχύει, όπως έδειξε και ο κύριος Γκέμπελς. Δεύτερον, οι επενδύσεις ε, είναι αδιάφορες και στο, στην αλλαγή των μισθών και στην, στο θέμα των κερδών. και τρίτον, οι ε, έχουν καταπέσει στην Ευρώπη λόγω της πολιτικής λιτότητας στην Ευρωζώνη. η εσωτερική ευρωπαϊκή ζήτηση έχει φτάσει στο μηδέν, έχει πέσει στον αδύρ. Ε, Αγαπητοί κύριοι, ε, έχετε κάποιες αμφιβολίες ε, για τις συστάσεις σας αυτές, θεωρείτε ότι κάπου έχετε κάνει λάθος. Ευχαριστώ. Τρία λεφτά η Κομισιόν ε, και εν συνεχεία το Δουνουτού. Όλοι. Ό,τι μπορεί σε τρία λεπτά να απαντήσεις. Ευχαριστώ Σάρον. Είναι μια πρόκληση. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιστρέψει αυτήν την τάση μαζί με την Ελλάδα. Αυτό το ρώτησαν και στους προηγούμενους γύρους, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα προηγουμένως. Η δουλειά που κάνει η Κομισιόν σε συμφωνία με την Ελλάδα και με τους εταίρους στην Τρόικα είναι η Ελλάδα να προχωρήσει με άμεση δράση για να υποστηρίξει την ε, νεολαία, να υπάρξει μια πρώτη εργασία, ώστε να αποκτήσουν ε, πείρα καταρχήν οι νέοι και επίσης να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες, ε, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις ουσιαστικά να επεκτείνουν τις μορφές μαθητείας, τις ευκαιρίες που δίνουν σε πτυχιούχους, σε νέους, για να προωθήσουν ε, την απασχόληση των νέων ε, με σκοπό να τους δώσουν κάποια προσόντα. Με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε την ε, απασχόληση των νέων. Ο Λάσλο Άντερ, ο συνάδελφός μου επίτροπος, προωθεί την προσπάθεια του Κοινωνικού Ταμείου ε, με δράσεις για να υποστηριχθούν οι νέοι ε, με μια ευρία δέσμη μέτρων, υποστήριξη νέων για να δημιουργήσουν ε, επιχειρήσεις, ευκαιρίες κατάρτισης, για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, να ενισχύσουν τους δεσμούς ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην εργασία. Αυτό είναι τμήμα του προγράμματος και συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα ούτω ώστε να ελαφρύνουμε ε, αυτό το βάρο τη μεγάλη ανεργία των νέων στην Ελλάδα. Μάθα τα μέτρα που σας είπα. Και βασίζομαι και στην ε, υποστήριξή σας γι' αυτό. Το άλλο θέμα που ακούστηκε, κύριε Πουπάκη, είναι αυτή η κοινωνική πλατφόρμα και ο κοινωνικό διάλογος που αναφέρατε. για αυτή την κοινωνική πλατφόρμα για την Ελλάδα με την ε, συμμετοχή των συνδικάτων, των οργανώσεων των εργοδοτών και των ε, διεθνών οργανισμών. Δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρξει κοινωνικός διάλογος τέτοιου είδους. Να συμπεριληφθούν και οι Έλληνες κοινωνικοί εταίροι, καθώς και οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις τους η εφαρμογή του προγράμματος δεν μπορεί να παραβιάσει τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα, ούτε το ενωσιακό δίκαιο. Η Κομισιόν είναι θεματοφύλακα της συνθήκης ε, και αναλαμβάνει τις ευθύνες της πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα πρέπει να σεβαστεί το ελληνικό σύνταγμα. Και οποιαδήποτε πολιτική συμφωνήσουμε με την ελληνική κυβέρνηση και υιοθετήσει το ελληνικό κοινοβούλιο, θα πρέπει να σεβαστεί το Σύνταγμα. Και αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με τόσα προβλέπει η ελληνική νομιτάξη. Κυρία Φερέρα, μίλησε για τις οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε κάποιες προϋποθέσεις, σε κάποιες εικασίες. Ε, για τις ε, μακροοικονομικές προβλέψεις, για το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και για τις ε, πολιτικές που προωθούνται στον τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Το 2010 και 2011, οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις στις οποίες βασιστήκαμε δεν ήταν σωστές. Ήταν, η πραγματικότητα ήταν χειρότερη. Αντίθετα από την περίπτωση της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, οι περισσότερες υποθέσεις στις οποίες βασιστήκαμε δεν ήταν σωστές. Πρέπει να τονίσω τη σημασία της αντιμετώπισης του προβλήματος του ασθενούς διοικητικού δυναμικού. Επίσης πρέπει να υπάρξει πολιτική ενότητα, ούτως ώστε να υπάρξει στήριξη ε, για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στη χώρα για την φορολογική μεταρρύθμιση. Κάτι που τόνισαν πολλοί ομιλητέ και τη σημασία τους. Θα πρέπει μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, το ελληνικό κοινοβούλιο, να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας για την φορολογική μεταρρύθμιση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Δεν είναι θέμα μόνο εισπράξεων και εσόδων από τους φόρους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για να επιτευχθούν βέβαια οι δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης αυτό και αποδοχής του προγράμματος. Για να υπάρξει αποδοχή θα πρέπει μαζί να βελτιώσουμε το δυναμικό της Ελλάδας να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσει το φορολογικό σύστημα, τόσο ώστε να είναι αποτελεσματικό και δίκαιο, ούτως ώστε οι πολίτες της Ελλάδας να πιστούν ότι φορολογία επιβάλλεται με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο. Τη βασική ευθύνη της φορολογικής μεταρρύθμισης την έχει η Ελλάδα και υποστηρίζουν την Ελλάδα τα μέλη του Δουνουτού, ε, η Task Force, αυτήν την προσπάθεια. Χαίρομαι από τη δέσμευση και την ταύτιση που υπάρχει, ε, όπως φαίνεται μέσα από τη σοβαρή συζήτηση. Ελπίζω να υπάρξει, να μετασχηματιστεί σε πραγματική βοήθεια και πραγματική στήριξη, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες σε αυτές τις φοβερές ε, προκλήσεις, ούτω ώστε να υπάρξουν ε, δουλειές και απασχόληση από τις μεταρρυθμίσεις θα χρειαστεί μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας, τη ελληνικής δημόσια διοίκηση και τη ελληνικής κοινωνίας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πολ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω με τον δημόσιο τομέα. Δεν αληθεύει ότι το πρόγραμμα επικεντρωνόταν πρώτα και κυρίαρχα όσον αφορά τα έσοδα, το σκέρος των εσόδων. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ήταν υπό πολύ οδυνηρές, σε οδυνηρές ε, ε, μειώσεις ε, των μισθών και των συντάξεων. Σημαντικές περικοπές και όσον αφορά και τις δαπάνες πέρα από τη μείωση συντάξεων και μισθών. Αληθεύει όμως ότι είδαμε κατά τη διάρκεια του 2011 ότι φτάσαμε το όριο. Το όριο του εφικτού και αυτού που μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά και την αύξηση της φορολογίας, του φορολογικού βάρους. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι επίσης φτάσαμε ένα σημείο και ένα όριο όπου δεν υπάρχουν πλέον εύκολες, εύκολα μέσα για τις δαπάνες που να είναι ισορροπημένα κοινωνικά, ισορροπημένα και δίκαια. Για να γίνει αυτό, αυτό θα απαιτήσει βαθύτατες, βαθιές μεταρρυθμίσεις, διαθωτικές μεταρρυθμίσεις και αυτό απαιτεί χρόνο, βάθος χρόνου για να επιτευχθεί. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Επίση όμω είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τρόικα εργάζεται με την ανάλυση και τη συζήτηση του συνολικού ελλείμματος και χρέους και του χαρτοφυλακίου που προτείνεται και οι ελληνικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα το κάνουν στο σκέλος των εσόδων ή των δαπανών. Και επειδή είδαμε ότι κάποιες από τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει ακόμα να γίνουν, γι' αυτό φαίνεται ότι υπήρχε συνένεση να περάσουμε στον τομέα των εσόδων. Αλλά με όλους που συζητήσαμε στην Ελλάδα, όλοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι φτάσαμε στο τέρμα της διαδρομής όσον αφορά την αύξηση των φόρων. Και υπάρχει συμφωνία ότι στο νέο πρόγραμμα, τουλάχιστον, η εξυγίαση, η εμπέδωση, η παγίωση πρέπει να γίνει όσον αφορά τις δαπάνες. Αυτό θα πάρει πολύ μεγάλο χρόνο γιατί θα απαιτήσει δυσχερείς, δυσχερέστατες διαθεωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Τώρα, Λάθος με ανέφεραν στα όσα είχα πει και δεν είναι σωστό το ότι είπα ότι δεν έχει ε, διοικητικό δυναμικό η Ελλάδα. Έχει κάποιους περιορισμούς όσον αφορά το διοικητικό δυναμικό της. Αυτό καθίσταται σαφές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πρώτα. Εμείς το μάθαμε αυτό, το είδαμε στην Ελλάδα. Τι κάνουμε. Συνθέτουμε και συσσωρεύουμε μεγάλο δυναμικό πραγματονομοσύνη για να βοηθήσουμε. Πέρσι είχαμε πάνω από 30 αποστολέ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε επαφέ με τι δημόσιε αρχέ στην Ελλάδα. Φυσικά αυτό δεν αποδίδει όπω εμεί προσδοκούσαμε και θέλαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χωρί ελπίδα η κατάσταση. Συνέχουμε, συνεχίζουμε να παρέχουμε αυτή την αρρωγή και ευελπιστούμε ότι το διοικητικό δυναμικό τη χώρα θα βελτιωθεί μακροπρόθεσμα. Τώρα για την διαχείριση το, του τομέα το, της εφορίας και των ε, φορολογικών θεμάτων. Συμφωνώ με τον Όλη Ρέν ότι έχει σημασία που είναι τεράστια η σπουδαιότητά της όσον αφορά το πρόγραμμα και τη συνέχιση του. Θα πήγαινα και πιο πέρα. Θα έλεγα κιόλα ότι δεν μπορώ να δω, βλέποντα τα αριθμητικά μεγέθη, του αριθμού, τα στοιχεία, και το ανέφερα αυτό προεισαγωγικά, δεν μπορώ να δω πώ μπορεί να διατηρήσει η Ελλάδα ένα σύστημα ευημερία όπου θα μπορεί κανεί να αναμένει από μια ευρωπαϊκή χώρα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποκατασταθεί ο έλεγχος των ε, ε, εσόδων χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ε, της ε, φοροδιαφυγής. Αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα της φοροδιαφυγής θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι υποχρεωμένη να περιορίζει τις κοινωνικές δαπάνες ε, και τις κοινωνικές, την, επένδυση στο κοινωνικό τομέα. Και αυτό θα είναι απαράδεκτο. Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει λοιπόν όσον αφορά τα φορολογικά θέματα και να αντιμετωπιστεί και η φοροδιαφυγή. Και όπως και όλοι οι ΡΕΝ και εγώ σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εγχείρημα η συζήτηση αυτή, η διαβούλευση αυτή, με όλες τις ερωτήσεις που δείχνουν ακαθόδη θέματα και ζητήματα. Σας διασφαλίζω ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση και εύρος ε, θεμάτων που εξετάζουμε. Πώς μπορεί να γίνει το ένα ή το άλλο. Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα με προσαρμογές που κάνουμε για να ανταποκριθούμε και ο, διάλογος το δείχνει είναι επικοδομητικό αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ο διάλογος είναι σημαντικός όπως θεωρείτε κι εσείς είναι ένας πρώτος διάλογος. Δεν πρέπει να είναι ο τελευταίος. Δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος. Σε όλα αυτά τα θέματα οικονομικών προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων αποκλείεται οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, οποιαδήποτε οργάνωση να τα καταφέρει εάν οι δράσεις της δεν είναι διαφανείς εάν δεν είναι αντικείμενο δημοκρατικής συζήτησης, εάν δεν αξιολογηθούν. Ακριβώς αυτό θέλαμε να εξασφαλίσουμε σήμερα. Από πλευράς μου καταλήγω σε τρία συμπεράσματα. Πρώτον, οι αξιολογήσεις δεν πήγαιναν όλες προς την ίδια Ανάλογα με την άποψη του καθενός, ανάλογα με την προέλευση του καθενός. Αυτή η προσπάθεια όμως είναι εκ των ονουκάνευ. Στο παρελθόν η Κομισιόν δεν ήθελε καν να δημοσιοποιήσει, θυμάμαι, το Memorandum of Understanding ε, που εφάρμοσε στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ τώρα για τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα που δείξατε. Καταλάβετε μας καλά. Υπάρχει ένα διακύβευμα για μας ε, δημοκρατικότητας. Ο κ. Ράσμουσεν είπε, ο κύριος Ράσμουσεν είπε ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του προγράμματος είναι η ικανότητα της ε, πολιτικής τάξης να ταυτιστεί με το πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ελαφρά με αυτό το σημείο. Νομίζω ότι δεν αρκεί η πολιτική τάξη να αποδεχτεί την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Εάν οι κοινωνικοί εταίροι, εάν οι Έλληνες πολίτες οι ίδιοι δεν πιστούν πλήρω για τη δικαιοσύνη του προγράμματο αυτού μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή, αποκλείεται να υπάρξει επιτυχία. Και το σχέδιο τη εναλλακτική λύση θα τεθεί τότε. Επομένω, το πρώτο βασικό θέμα είναι η δημοκρατία, η διαφάνεια, η νομιμότητα αυτού του προγράμματο. Και το εγχείρημα που κάνουμε σήμερα μα διδάσκει κάποια πράγματα. Ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να κάνετε αυτή την προσπάθεια πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, πριν εφαρμοστεί το πρόγραμμα και πριν προσδιοριστεί από τις αρχές ε, που το καθορίζουν. Το δεύτερο συμπέρασμα, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όταν κοιτάμε την άποψη της Τρόικα, την προσέγγιση της Τρόικα, Βλέπουμε μια προσέγγιση του κέντρου προς την περιφέρεια. Αντιμετωπίζουμε το ελληνικό ζήτημα χωρίς να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα θέματα που μπαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν έκανε την αξιολόγηση των 10 ετών λειτουργίας της Ευρωζώνης, είχε πει ότι το α και το ω του προβλήματος της ε, λειτουργίας της ζώνης ευρώ ήταν το θέμα των εσωτερικών ανισορροπιών της Ευρωζώνης ξέρω πολύ καλά ότι είναι η εντολή σα, ότι είναι η αποστολή σα. Εσεί είστε μέσα στην κατάσταση. Ε, αντιμετωπίζετε από μέσα το ελληνικό πρόβλημα. Αλλά εμεί έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε μέσα σε ένα τσολίνα ή μέσα σε ένα τούνελ, δεν ξέρω πώ να το πω, όπου μόνο η δική σα άποψη στο ελληνικό ζήτημα επιλύει, το επιλύει κατά ανάγκη. Οποιοδήποτε παρατηρητή που σκέφτεται ε, λέει ότι ανεξάρτητα από τη δική σα οπτική Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και άλλες οπτικές γωνίες. Ο Ζαν Πολ λέει ότι η κρίση της ε, Ελλάδας δεν είναι η κρίση της Ευρωζώνης. Αλλά αν η Ευρωζώνη είχε λειτουργήσει τέλεια, δεν θα υπήρχε και η ελληνική κρίση στο κάτω-κάτω. Όλες αυτές οι σχέσεις, οι διασυνδέσεις, ε, είμαστε συνυπεύθυνοι, ε, υπάρχει αλληλεγγύη, έχουμε το ίδιο νόμισμα. Ε, υπάρχει λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής ε, Ένωσης. Ε, η οποία δεν λειτουργεί απόλυτα καλά. Υπάρχουν ανισορροπίες και ένα από τα συμπτώματα αυτών των ανισορροπιών είναι η Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι αυτό λείπει από την άποψή σας, από την οπτική σας γωνία για το ελληνικό ζήτημα. Και το τελευταίο συμπέρασμα ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Κύριε Ρεν, στο τέλος, στο τέλος μιλήσατε για δικαιοσύνη, fairness. Κανένας δεν μίλησε όμως για την κοινωνική δικαιοσύνη. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι που δεν έφερα ένα δώρο σε καθένα από εσά. το βιβλίο του Βίλκινσον που λέει γιατί η, η δίκαιη κοινωνία είναι καλύτερη για όλους. Γιατί η οικονομική αποτελεσματικότητα βασίζεται και στην κοινωνική, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι η άποψη τη επιτροπή Απασχόληση ε, είναι να σας πω ε, τις απόψεις του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας. Ε, θα πρέπει να λυθούν οι υπόψεις στην αξιολόγησή σας. Θεωρούν ότι αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπου θεωρείται ότι το μοναδίο κόστος εργασίας είναι μία βασική παράμετρος, είναι μια βασική παράμετρος, βασικη παραμετρο όχι μόνη για την διόρθωση του ελληνικού προβλήματο. Δεν θέλω να πω περισσότερα σε αυτή τη φάση. Θέλω απλώ να σε ευχαριστήσω εν ονόματι και των δύο επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών, εν ονόματι ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την προσπάθεια. Σας ξαναδίνουμε ραντεβού για άλλες αξιολογήσει. γιατί αποκλείεται να μείνουμε εδώ σε αυτές τις διαπιστώσεις. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σήμερα.